Your colleagues. Um, we can start our... συνάδελφοι, θα αρχίσουμε τη συνεδρίασή μας για το απόγευμα. Καλωσορίζω την Έλκια Κιόνιχ. Όπως ξέρετε είναι πρόεδρος του ενιαίου οργανισμού εξυγένσης την είχαμε κοντά μας στις 20 Μαρτίου. Σήμερα θα μας παρουσιάσει την ετήσια έκθεση του οργανισμού της για το 2017. Όταν ήρθε εδώ πριν από ένα χρόνο, το SRB είχε ε, περάσει από την πρώτη κρίση της ε, λειτουργίας του και χαιρόμαστε που τους τελευταίους μήνες, παρόλες τις δυσχέρειες που υπάρχουν, δεν είναι τόσο Εντυπωσιακέ εξελίξεις. Υπάρχουν σημαντικές ε, εξελίξεις όμως, ιδιαίτερα το Eurogroup και η συνάντηση κορυφή ε, του Ιουνίου. Όπως ξέρετε, υπάρχει συμφωνία που λέει ότι το ESM θα είναι ο ίστατος μηχανισμός ασφαλείας. Δεν είναι καινούριο, αλλά πρέπει να καθοριστούν οι λεπτομέρειες λειτουργίας και τα θέματα διακυβέρνησης που μπορεί να καθορίσουν τη διαφορά ανάμεσα σε έναν μηχανισμό ίστα της ασφαλείας και ένα πρόγραμμα. Σήμερα ξεκινήσαμε τον τριμερή διάλογο για την αναθεώρηση των κανονισμών BRD και SRM. Σημαντική λοιπόν ημερομηνία για τις διαδικασίες εξυγίανσης θα έχουμε λοιπόν πιστεύω πολύ ενδιαφέροντα θέματα να συζητήσουμε. Οπότε έλκε, σου δίνω το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, Αξιότιμα μέλη. Δεν ξέρω, είμαι το τελευταίο εμπόδιο μεταξύ της δουλειάς σας και των θερνών διακοπών, αλλά ξέρω ότι θα πάτε και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως πάντα, είναι μεγάλη χαρά η συμμετοχή μου και θα κάνω ό,τι μπορώ για να απαντήσω στις ερωτήσεις σας. Με καλέσατε σήμερα για να σας παρουσιάσω την ετήσια έκθεση δραστηριότητας για το 2017. Αλλά επειδή το 2017 ε, μοιάζει να έχει λήξει εδώ και πολύ καιρό, θα αξιοποιήσω την ευκαιρία για να κοιτάξω και τα άλλα τρέχοντα θέματα και ορισμένα θέματα που ήδη αναφέρατε. Για να σχολιάσω την ε, υποεξέλιξη, υποεξέλιξη συζήτηση για το πακέτο μείωσης των κινδύνων και ορισμένα άλλα θέματα. Οπότε, ξεκινάω. Όπως είπατε, πέρυσι τέτοια εποχή, συγκεκριμένα στις 6 Ιουνίου, το SRB αντιμετώπισε την πρώτη της ε, υπόθεση, την εξυγένση της Banco Popular στην Ισπανία. Ήταν ε, πολύ σημαντικό γεγονός. Απέδειξε, γιατί το ξεχνάμε πολύ συχνά, ότι ο οργανισμός μας μπορεί να εφαρμόσει τους ε, ισχύοντες κανόνες και να εκτελέσει την εντολή της, ούτως ώστε να υπάρξει μια διατεταγμένη εξυγένση με ελάχιστη επίπτωση στην πραγματική οικονομία, το χρηματοπιστωτικό σύστημα και τα δημοσιονομικά του αντιστοίχου κράτους μέλους και ευρύτερα. Πολλή δουλειά όμως γίνεται για τα θέματα αυτά και θα επανέλθω στην περίπτωση της Banco Popular το 18. Αλλά πιστεύω ότι απέδειξε καθαρά ότι η εξυγίανση μπορεί να διασφαλίσει την ε, οικονομική σταθερότητα και σε αυτή την περίπτωση την ε, εξασφάλισε. Το 17 επίσης ε, προχωρήσαμε πολύ και τις δραστηριότητες μας για την εξυγένση των ομίλων τραπεζών υπό την επιτήρησή μας. Έτσι λοιπόν διασφαλίσαμε ότι οι τράπεζες είναι πραγματικά εξυγιάνσιμες. Αυτό είναι ένα πολιτές πρόγραμμα, αλλά κάναμε βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Και στο τέλος του 2017 δημοσίευσαμε, δημοσίευσαμε την πολιτική μας για τα MREL, που έδωσε και στις τράπεζες και τους πιστωτές, σε όλους τους εμπλεκομένους, σαφή κατεύθυνση για το τι θέλουμε να γίνει τα επόμενα χρόνια από τις τράπεζες. Επίσης, είχαμε και συμπροματικές πολιτικές και κατευθυντήρες γραμμές που δημοσιεύθηκαν και είπαμε και ε, θέσαμε τους πρώτους targets MRL σε συνολικό επίπεδο για τις πιο σημαντικές ε, ομάδες τραπεζών. Δηλαδή για 80% περίπου των ενεργητικών των τραπεζών στην ε, Τραπεζική Ένωση και δώσαμε και πληροφορίες για στόχους για τις άλλες τράπεζες και σας διαβεβαιώνω ότι το καταλαβαίνει ο κλάδος απόλυτα αυτό. Οπότε, εάν ξέρεις ε, προς τα που πάει η κατεύθυνση, δεν χρειάζεται να περιμένεις για δεσμευτικούς στόχους, ε, εφόσον είναι ευνοϊκές και οι αγορές. Επίσης, συνεχίσαμε την περισσότερη προσπάθεια για να λειτουργήσει το ταμείο, το ενιαίο ταμείο ε, εξυγένσης ε, στις τέλους Ιουνίου οι εθνικές ε, ρυθμιστικές αρχές είχαν ήδη εμβάσει 60 συμβολές 7,5 δισεκατομμύρια στο SRF το οποίο σημαίνει ότι τώρα έχει περίπου 25 δισεκατομμύρια. Και σημειώνω ότι εξεπλάγει κάπως ο κλάδος γιατί σε σχέση με πέρυσι, φέτος αυξήθηκαν οι συνεισφορέ κατά 3%. Αλλά αυτό οφείλεται στο θετικό γεγονός ότι αυξήθηκαν κατά περίπου 3% οι καταθέσεις πέρυσι. Οπότε για να επιτύχουμε το στόχο του 1% καλυπτωμένων καταθέσεων, είχαμε την ετήσια συνεισφορά και ε, είμαστε αρκετά σίγουροι ότι ο τελικός στόχος για το Ταμείο θα είναι πολύ πάνω από την αρχική πρόβλεψη 55 δις. Βέβαια πρέπει να κάνουμε και τα εσωτερικά μας καθήκοντα. Τώρα έχουμε περίπου 300 ε, εργαζομένους και μόνιμους και προσωρινούς. Δηλαδή φτάσαμε περίπου, ε, θα φτάσουμε μάλλον, στο επίπεδο της ε, του προσωπικού που θα θέλαμε για το τέλος του χρόνου. Η εργασία μας φυσικά δεν σταματάει ποτέ. Αλλά να αναφερθώ στο, στην Banco Popular. Στις 30 Ιουνίου ανακοινώσαμε ότι είχαμε πάρει την ε, τελική αποτίμηση και την έκθεση που έλεγε ότι ε, θα είχαν ε, υποστεί καλύτερη μεταχείριση οι πελάτες και οι πιστωτές αν είχε εξηγιανθεί η τράπεζα με ε, τις κανονικές διαδικασίες ε, Και έχουμε μία προπαρασκευαστική δράση και μία μη εμπιστευτική ε, εκδοχή της ε, έκθεσης της εξολόγησης 3. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν τη διαδικασία εγγραφής για το δικαίωμα να ακουστεί η φωνή των πάντων στις αρχές Αυγούστου. Έτσι και οι μέτοχοι και οι πιστωτές και οι πελάτες που εθίγησαν θα ε, μπορέσουν να ασκήσουν το δικαιωμά τους αν το επιθυμούν, να το δηλώσουν δηλαδή και ξέρουμε ότι όταν ε, ξεκινάει η διαδικασία αρχές Αυγούστου ε, είναι βέβαια στη μέση των διακοπών. Θα συνεχιστεί λοιπόν μέχρι το Σεπτέμβριο για να έχουν όλη τη δυνατότητα να εγγραφούν. Αυτή και η προπαρασκευαστική εργασία και η μη εμπιστευτική εκδοχή της ε, αποτίμησης 3 θα είναι έτοιμη μέχρι τότε και σε μια δεύτερη φάση τα άτομα των οποίων ελέγχθηκε η επιλεξιμότητα από το SRB θα μπορέσουν να υποβάλουν τα σχόλιά τους για την προπαρασκευαστική μας ενέργεια για θα αποζημιωθούν με βάση την έκθεση που κάναμε οι μέτοχοι και οι πιστωτέ. Αυτό θα γίνει όταν θα ολοκληρωθεί η διαδικασία καταγραφής. Θα πάρει κάποιο χρόνο. Αλλά είναι προς το συμφέρον της χρηστής ε, διοίκηση. Και είναι αναγκαίο να γίνει κάτι τέτοιο πριν λάβουμε την τελική απόφαση. Τώρα να επανέλθω στην κανονική εργασία μας. Έχουμε πάντα κατά νου ότι ο προγραμματισμός της εξυγίανση είναι πολυετής προσπάθεια. Για το 2018 έχουμε ήδη εργαστεί και θα εργαστούμε για να ολοκληρώσουμε τα σχέδια εξυγίανση για όλες τις τράπεζες υπό τον έλεγχό μας. Και θα θέσουμε λοιπόν στόχους MRL για όλες τις τράπεζες. Αλλά όπως έχω επανειλημμένα πει, αυτό θα φτάσει μέχρι το 2020 μέχρι να ολοκληρωθεί συνολικά με βάση το πολιτές πρόγραμμα εργασιών μας. Επιπλέον, ασχολούμεθα με τις ε, πολιτικές γενικότερα. Μία συγκεκριμένη είναι αυτή που δημοσίευσαμε τον Μάιο για τις κρίσιμες λειτουργίες. Δεν ξέρω αν το ξέρετε, αλλά το συζητήσαμε και το εκλεπτήναμε ήδη από τις αρχές του 2016 και ωφελήθηκε από πολλά διδάγματα από τον πρώτο κύκλο ε, προγραμματισμού εξυγίανσης. Είναι ουσιώδες ε, στοιχείο για να καθορίζουμε εάν μια προβληματική τράπεζα πρέπει να εξυγιανθεί ή εάν θα υπάρξει διαδικασία αφαιρεγγιότητας. Όταν ξεκινήσαμε είχαμε τράπεζες που είχαν 100 κρίσιμες λειτουργίες, μικρές. Και Άλλοι οργανισμοί δεν θεωρούσαν ότι έχουν κανένα, καμία κρίσιμη λειτουργία. Προσπαθήσαμε να αναρμονίσουμε την κατάσταση. Τα δημοσιεύσαμε αυτά και ελπίζουμε έτσι να παράσχουμε διαφάνεια και στις τράπεζες και να διασφαλίσουμε τη συνέπεια στον καθορισμό, τον εντοπισμό μάλλον, των κρισίμων <clears throat> λειτουργιών. Και έχει γίνει θετικά δεκτό. Επίσης υπάρχει πρόοδος για να ολοκληρώσουμε τις δικές μας τι εσωτερικέ γραμμές για τι ομάδε μα. Για το πώ θα αντιμετωπίσουν το όργανο, την τράπεζα γέφυρα, για παράδειγμα την ε, διάσωση με την συμμετοχή των καταθετών και τη διαδικασία διαχωρισμού των στοιχείων ενεργητικού και όλα αυτά νομίζω ότι θα τελειώσουν στο τέλος του ε, φινοπόρου και θα υπάρξει ένα δημόσιο εγχειρίδιο. Και έχει να κάνει πολύ με το διάλογο που έχουμε με τον κλάδο, με τις τράπεζες και χωρισμένα, ούτω ώστε να είναι προσαρμοσμένα στι ανάγκε του. Θα μπορούσα να μιλήσω για πολλά για την αποτίμηση, τη ρευστότητα, τη χρηματοδότηση κτλ. Αλλά το σημαντικό είναι ότι παρά τα σχέδια εξυγίανση ε, που είναι ακόμη από εξέλιξη, καμία τράπεζα που έχει υπεύθυνη διοίκηση δεν θα πρέπει να περιμένει να του στείλουμε συγκεκριμένε εντολέ. Οι τράπεζε ξέρουν πολύ καλά τι πρέπει να κάνουν. Του έχουμε σαφώ ε, ενημερώσει για τις απαιτήσει μας και για το πρόγραμμα εργασιών για το 2018, το οποίο είναι προσαρμοσμένο επί μέτρο σε κάθε πιστοτικό ίδρυμα. Και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Και θα παρακολουθούμε και τη συνέχιση. Γιατί είτε οι, τράπεζε οι τράπεζες πρέπει να γίνουν από μόνος τους εξι... και εμείς να τις πιέσουμε. Οι τράπεζες γνωρίζουν την κατεύθυνση της πορείας μας και νομίζω ότι μπορούν να εργαστούν. Αυτό ισχύει και για το MREL. Και τα καλά νέα είναι ότι σημειώνεται πρόοδος από αυτού. Τώρα, με συγχωρείτε ξέρω ότι μακρηγορώ, θέλω να παρέσω τώρα στο πακέτο για τη μείωση των κινδύνων, κάτι που με ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Και ιδιαίτερα την αναθεώρηση του BRRD και του SRMR, νομίζω ότι έχουμε μπει σε αποφασιστική φάση. Τώρα που και το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενέκριναν τις θέσεις τους. Ελπίζω λοιπόν ότι θα προχωρήσουμε γρήγορα και θα καταλήξουμε σε μια καλή συμφωνία όσο ταχύτερα υπάρξει σαφήνεια για τις δραστηριότητές μας και για τους ε, οργανισμούς που δρούν στην αγορά, τόσο το καλύτερο. Γιατί βεβαίως ε, θα αναθεωρηθεί μια οδηγία και μέχρι να μεταφερθεί στα εθνικά δίκαια θα πάρει χρόνο. Τώρα, μερικές διατάξεις. Ένα τομέα όπου μας ε, ικανοποιεί ιδιαίτερα η συμβολή του Κοινοβουλίου είναι η απλούστευση. Όσο και αν θέλετε να το βελτιώσετε, αλλά όλα αυτά θα βοηθήσουν μόνο τους δικηγόρους που θα αρχίσουν να κοιτάνε τις λεπτομέρειες. Η, απλότητα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό. Και για ένα άλλο λόγο. Γιατί μόνο έτσι υπάρχει αναγκαία διαφάνεια και προβληψιμότητα για τα πιστοτικά ιδρύματα, για τους επενδυτές και νομίζω και για το κοινό γενικότερα. Επίσης πιστεύουμε ότι το ποσοστό των MREL πρέπει να συνδυάζεται με την στρατηγική εξυγένση κάθε πιστοτικού ιδρύματος. Είναι το μέσο που είναι αναγκαίο για να είναι εξυγιάνσιμη μια τράπεζα Αντιμετωπίζοντα τις δυσχέρειε. Οπότε, είμαστε υπέρ μια σημαντικής ε, ε, ενός σημαντικού τμήματος ε, δευτερευόντων MRL. Τώρα ο τρόπος που θα γίνει ταξινόμηση θα πρέπει να βελτιώσει την την ε, εξηγενσιμότητα και να τηρείται η αρχή του ότι κανένας πιστωτής δεν θα πρέπει να ε, καταλήξει χειρότερα για να μπορούμε να λάβουμε δράση εξυγίανσης με, διαφάνεια ούτω ώστε οι επενδυτέ να μην ισχυριστούν μετά ότι δεν ήξεραν τι είχαν αγοράσει. Αλλά μην με παρανοήσετε. Δεν λέω ότι μόνο τα δευτερεύοντα μέσα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την, ε, την ε, διάσωση με συμμετοχή των ε, καταθετών και μετόχων, αλλά πρέπει να είναι καθαρά τα πράγματα. Δυστυχώς το κείμενο του Συμβουλίου είναι πιο κοντά στις δικές μας απόψεις. Όσον αφορά τα δευτερεύοντα MRL. Το άλλο είναι να υπάρχει δυνατότητα επιλογής για την ποιότητα και την ποσότητα. Και κάτι άλλο που είναι πολύ σημαντικό και για μας, αλλά και για σας από ό,τι καταλαβαίνω, το επιχείρημα ότι πρέπει να υπάρχουν εσωτερικά μέσα MREL είναι απόλυτα σαφές. Αλλά πρέπει να επιτηρούνται προσεκτικά. Ότι ο καθορισμός των MREL πρέπει να είναι τμήμα της στρατηγικής εξυγίανσης που να εντάσσεται στη στρατηγική εξυγίανση του ομίλου πιστοτικών ιδρυμάτων. Δηλαδή, να μην αντιτίθενται αυτή η προσπάθεια στην προσπάθεια να μην δημιουργούνται επιπλέον φραγμοί. Τέλος, καλωσορίζουμε το νέο ε, εργαλείο διακοπής, Moratorium Tool, που μπορεί να εφαρμοστεί εάν μια τράπεζα κινδυνεύει να καταρρεύσει. Αλλά δεν θα ήθελα να αξιοποιήσουμε τις ε, δυνατότητες ε, αναβολής μόνο για 10 μέρες. Εγώ πιστεύω ότι δεν είναι αναγκαίο αυτό. Θα μπορούσε μάλιστα να είναι και αντιπαραγωγικό, να έχει τα αντίθετα αποτελέσματα. Λοιπόν, να σταματήσω εδώ και ευχαρίστω θα συμβάλλουμε στον τριμερή διάλογο, αν μας το ζητήσετε, και ίσως να το κάνουμε και αν δεν μας το ζητήσετε, απλώς να σας στείλουμε τις απόψεις μας. Άλλα θέματα τα αναφέρατε, αναφέρατε ένα, εγώ θα ξεκινήσω με ένα άλλο. Έχω την εντύπωση ότι δυστυχώς το έντις το σύστημα εγγύησης των καταθέσεων δεν έχει προχωρήσει σημαντικά τον τελευταίο χρόνο, αλλά πιστεύουμε ότι το ΕΝΤΙΣ ως τρίτος πυλώνας της Τραπεζικής Ένωσης πρέπει να γίνει πραγματικότητα. Και βασιζόμεθα σε εσά και στην ε, Προεδρία του Συμβουλίου να μην το αφήσει κατά μέρο εντελώ. Είναι πάντα θέμα χρόνου και προγραμματισμού, αλλά θα πρέπει να μείνει επιτάπητος. Το πρόσφατο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για άλλη μια φορά απεκάλυψε ότι υπάρχει πολιτική συνένεση για την ανάγκη για ένα κοινό μηχανισμό ασφαλείας, ένα common backstop. Οπότε τονίζω ότι πρέπει να συμφωνήσετε στα οργανωτικά μέτρα από αυτού. Είπατε ότι δεν είναι ένα backstop αναχώρα, είναι ένα backstop για την αρχή εξυγένσης και σε περίπτωση ανάγκης η συμπληρωματική βοήθεια, ελπίζω ποτέ να μην τη η συμπληρωματική βοήθεια του backstop θα πρέπει να μπορεί να χορηγηθεί χωρί καθυστέρηση. Το γεγονό ότι το backstop είναι δημοσιονομικά ουδέτερο και χρησιμοποιείται μόνο ω ίστατη καταφυγή διασφαλίζει ότι οι φορολογούμενοι θα προστατευτούν. Αλλά είναι επίση σημαντικό να γνωρίζουμε ότι δεν μπορούμε να αποφασίσουμε για μια εξυγένση αν δεν έχουμε σαφήνεια για το πώς θα την ε, εφαρμόσουμε. Τέλος, και το έχω ξαναπεί, η χρηματοδότηση της εξυγίανσης είναι ανοιχτό θέμα γιατί πρέπει να γνωρίζουμε ότι δεν επιλύεται με το backstop στο SRF. Οι διαστάσεις δεν θα επαρκούσαν για να δώσουν επαρκή ρευστότητα αν ε, καταρρεύσει μια πολύ μεγάλη τράπεζα. Πρέπει λοιπόν να συνεχίσουμε να διερευνούμε εναλλακτικέ επιλογέ, ιδιαίτερα σε συνεργασία με τι Εθνικέ Κεντρικέ Τράπεζε και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Και τέλο, σα υπενθυμίζω και το έχω ξαναπεί, οι διαδικασίε αφαιρεγκαιότητα είναι αποκλειστικά θέματα εθνική νομοθεσία. Και γι' αυτό υπάρχει η περίπτωση της EBLB, αλλά και άλλες περιπτώσεις υπάρχουν, γι' αυτό δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε την προσπάθεια για να υπάρξει ευρωπαϊκή λύση, εάν όχι συνολικά για την αφαιρεκαιότητα, αλλά τουλάχιστον για την τραπεζική της πτυχή. Έχουμε πολλά προγράμματα, πολλές πρωτοβουλίες για να ενισχύσουμε το ευρώ και να καταλήξω θετικά. Είμαστε δεθυμένοι τώρα που ε, ο ήλιος είναι καλή οικονομική κατάσταση, να ολοκληρώσουμε το τραπεζικό πακέτο, να δημιουργήσουμε το backstop και όσο μπορούμε να βοηθήσουμε, ευχαρίστω να βοηθήσουμε. Και με συγχωρείτε αν ξεπέρασα τον χρόνο. Σας ευχαριστώ πολύ. Είχατε πολλά στοιχεία να μας δώσετε, οπότε ήταν λογικό να υπερβείτε το χρόνο, γιατί είχατε πολλές πληροφορίες να μας δώσετε και νομίζω ότι έπρεπε να σας ακούσουμε. Έχει πολύ μεγάλη σημασία επί της ουσίας βεβαίως και η διαδικασία έχει μεγάλη σημασία για το κοινό και χαιρόμαστε ιδιαίτερα που μας δώσατε πληροφορίες. Ο Μπουρχάλτ Μπάλτς έχει το λόγο από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κυρία Κόνιχη. Εδώ εκπροσωπούμε τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και όχι μόνο τα κρατημέλη. Αλλά όποιος έχει έτσι αρμοδιότητα ευρωπαϊκή, προφανώς και ενδιαφέρεται ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις ευλέψεις μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας από το Ιουνίου. Τις παρακολουθήσαμε λοιπόν ε, με προσοχή σε ό,τι αφορά τον οδικό αυτό χάρτη, σε ό,τι αφορά την ε, Τραπεζική Ένωση, μεταξύ άλλων ε, και τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και το πώς θα εξελιχθούν. Είναι ενδιαφέρον ότι οι δύο τόσο μεγάλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, σε ό,τι αφορά το, τα δευτερεύοντα MRL δεν τοποθετούνται πάντα με τον ίδιο τρόπο. Και τώρα, σε ό,τι αφορά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, αναφέρεται και παραθέτω από το UMPL, υποστηρίζεται η πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η πρόταση της ε, ECP για τα υφιστάμενα MPL, ε, θα πρέπει να έχουμε το 5% ε, ακαθάριστο και 2,5% καθαρά MPL, μη εξυπηρετούμενα δάνεια για όλε τι τράπεζε τέλος παράθεσης. Αυτό είναι θετικό σήμα και ένδειξη για την περαιτέρω μείωση του κινδύνου σε ό,τι αφορά την Τραπεζική Ένωση στην Ευρωζώνη. Η ερώτηση που έχω να σα απευθύνω είναι η εξή. Πώς το αξιολογείτε αυτό. Και κατά δεύτερον, στο τέλο τη παρέμβαση σα, μα είπατε κάποια ενδιαφέροντα σχόλια για το θέμα αυτό. Θέλω να εμβαθύνουμε, αν μου επιτρέπετε. Νομίζω ότι αντιληφθήκαμε ότι μέχρι τα τέλη του χρόνου σκοπός μας είναι να, αναπτυχθεί, να αναπτυχθούν κριτήρια για τον μηχανισμό ασφάλειας, τον backstop για την ανακεφαλαίωση ε, το ERSM, να την εγκαταστήσει ουσιαστικά. Αυτή η άμεση λοιπόν ανακεφαλαιοποίηση συνείδητα ε, και με πιο αυστηρούς ε, όρους. Αν τώρα το backstop πάρει άλλη τροπή. Θεωρώ ότι θα πρέπει να διατηρηθεί η αιρεσιμότητα. Και ποιε ε, είναι οι συνθήκε, ποιοι είναι οι όροι που θεωρείτε ότι είναι πιο σημαντικοί, προκειμένου αυτό το backstop, ο μηχανισμό ασφάλεια, να διαμορφωθεί σε ένα αποτελεσματικό εργαλείο, το οποίο θα είναι και ευρέω αποδεκτό. Ευχαριστώ. 2,5% και 5% στο γαλλογερμανικό έγγραφο. Αυτό το ποσοστό αναφέρθηκε, έτσι δεν είναι όχι στο έγγραφο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Η απάντηση της κυρίας Κονέχια για να μιλήσουμε για το έγγραφο αυτό της Γαλλίας και της Γερμανίας. Το εξέτασα με προσοχή, γιατί προφανώς θα πρέπει να σημειωθεί μια πρόοδος και νομίζω ότι περιλάμβανε πάρα πολλά στοιχεία τα οποία κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση. Σε ό,τι αφορά τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, νομίζω ότι κανείς δεν διαφωνεί ότι θα πρέπει να κινηθούμε προς τα εμπρός και νομίζω ότι και το έγγραφο αναφέρει ότι έχει σημειωθεί πρόοδος ήδη. Εγώ πάντα είμαι διστακτική όταν αναφέρονται ε, αριθμητικά στοιχεία σε ό,τι αφορά το 2,4%, το 2,5%, το 5%. Νομίζω ότι ο συνολικός στόχος όμως της μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων είναι αδιαμφισβήτητος και εκτιμώ τις προσπάθειες που καταβάλει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εγώ όπως σας είπα, πάντα ε, διστάζω όταν μιλάμε για ένα συγκεκριμένο αριθμητικό στοιχείο. Δεν ξέρω κατά πόσο στέκει, δεν ξέρω κατά πόσο ε, είναι σωστό. Είναι η άποψή μου αυτή, αυτή και ζητήσατε για τον backstop, ε, για τον ανασταλτικό αυτό μηχανισμό. Έχουμε την εργαλειοθήκη ESM, όπου έχουμε την άμεση ανακεφαλοποιήσει με αυστηρή ρεσιμότητα. Το θέμα της ρεσιμότητας στο backstop είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, γιατί προφανώς ο μηχανισμός ασφάλειας του backstop είναι ένας μηχανισμός δανειοδότησης στην αρχή εξυγίανσης. Δεν είναι ένα πρόβλημα το οποίο μεταφέρεται σε μια χώρα. Άρα, εγώ θεωρώ ότι ο μηχανισμός ασφάλειας είναι προφανώ. Ε, Όποιο σου δίνει μια πίστοση πρέπει να ξέρει ότι μπορεί να επιστρέψει το δάνειο αυτό. Αλλά δεν είναι δυνατόν να υπάρχει και δεύτερο επίπεδο αιρεσιμότητα ε, στο πρόγραμμα εξυγίανση. Εμεί ω ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανση θα χρησιμοποιήσουμε μόνο το δικό μα ε, ταμείο. Και αυτό θα είναι πρώτο. Όπου πιστεύουμε ακράδαντα ότι υπάρχει μια βιώσιμη λύση για κάποιο πρόβλημα. Άρα το Ταμείο θα πρέπει να ακολουθήσει την ίδια αιρεσιμότητα. Δυσκολεύομαι να φανταστώ μια δεύτερη φάση, ένα δεύτερο επίπεδο αμφισβήτησης μιας απόφασης εξυγένσης. Για μένα τα πράγματα είναι απλά. Έχουμε ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα και Συμφωνώ απόλυτα ότι όπως και οι τράπεζες και εμείς θέλουμε να ξέρουμε κατά πόσο θα πάρουμε τα λεφτά μας πίσω. Μέχρι εκεί όμως, γιατί ιδάλλως δημιουργούμε μια δεύτερη αρχή εξηγένσης. Συγγνώμη αν τα είπα πολύ καθαρά και εξάστερα. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Η κυρία euh, très... Σας ευχαριστώ για αυτά τα σαφέστατα λόγια για το πόσο περνάμε σε, από μία πιστοτική γραμμή σε μία άλλη μέσα στα πλαίσια της ερεσιμότητας που δεν θίξατε, γιατί ο συνάδελφος μίλησε για οικονομική ερεσιμότητα, αλλά υπάρχει και η διακυβερνητική. Δεν αφορά ίσως αρμοδιότητά σας, αλλά το ζήτημα είναι πώς έχει αυτή η διάρθρωση με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας δεν είναι απλά τα πράγματα. Ε, χαίρομαι που σας προβληματίζουν τα στοιχεία, αλλά υπάρχουν ορισμένα στοιχεία στα οποία είσαστε σαφέστατε. Υπάρχει ένα θέμα που μας απασχολεί εδώ στο Κοινοβούλιο, τα διδάγματα που θα πρέπει να αντλήσουμε από την περίπτωση της Λετωνίας και ιδιαίτερα της κατηγορίες διαφθοράς σε σχέση με τον πρώην διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας, ο οποίος παρετήθηκε. Βεβαίως η ΕΚΤ έχει κάνει προσφυγή στο δικαστήριο. Είναι μια διαδικασία κάπως αμήχανη, αλλά αυτό δείχνει ότι υπάρχει ένα κενό στην ομοθεσία γιατί είναι δύσκολο εάν κάποιος έχει προβεί σε τέτοιες πράξεις να μην διωχθεί, γιατί φυσικά έχει μεγάλη σημασία και η φήμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, γιατί ένα μέλος του Συμβουλίου θα μπορούσε να διωχθεί για διαφθορά. Αναρτιέμαι ως πολίτης, αλλά ε, θα ήθελα να πω ότι ίσως θα πρέπει να αλλάξει και το καθεστώς της ΕΚΤ. Και τώρα προς εσάς, σε σχέση με τα μέσα που διαθέτουμε για την νομιμοποίηση από παράνομα έσοδα και μετά από την περίπτωση της Λετωνίας, υπάρχουν συγκεκριμένες ε, διατάξεις ε, τύπου BRD, αλλά θα θέλαμε να μας πείτε τι μπορεί να γίνει ως προς την εξυγίανση τέτοιων τραπεζών, γιατί είδαμε ότι στην περίπτωση της Λετωνίας ότι μία τέτοια κατηγορία μπορεί να ενέχει και τον κίνδυνο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Θα ήθελα να σταθώ στο μηχανισμό ασφαλείας. Γνωρίζω πώς ε, κινείται ε, το ESM και αυτό ε, ίσως έχει να κάνει με μία αντίφαση με την δράση της, του ΕΣΕ. E δηλαδή δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να λάβουμε μία απόφαση εξυγίανσης ε, τάχιστα εμείς. Ε, σε αυτή την περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο του ESM μπορεί να ζητήσει μία πιστοτική γραμμή και όπως σας είπα, σε μία τέτοια περίπτωση ίσως θα πρέπει να ληφθεί άμεσα μία απόφαση, μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο δηλαδή και όταν αποφασίσουμε εμείς θα περάσουμε την απόφαση στην Επιτροπή, στο Συμβούλιο και ούτω καθεξής για να αρχίσει η διαδικασία έγκρισης. Η απόφαση αυτή δεν μπορεί να ληφθεί χωρίς να υπάρχει ασφάλεια ότι τα χρήματα είναι διαθέσιμα. Αυτό είναι ένα θέμα προς επίλυση, ελπίζω όμως να γίνει κατανοητό από όλους. Περιμένω λοιπόν την εργασία της Task Force να δούμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα αυτό. Ως προς τη Λετωνία, επειδή το θέμα δεν σχετίζεται με την εργασία του Συμβουλίου, του ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης, το θέμα της ε, διακυβερνητικής διάρθρωσης και της κατηγορίες κατά του διοικητή της ε, Λετονικής Κεντρικής Τράπεζας και τι σημαίνει αυτό για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Είναι πολύ δύσκολο να δούμε ποιος έχει δίκιο και ποιος σφάλει. Αλλά Εδώ με ρωτάτε ως πολίτη. Εάν ένας διοικητής δεν ασκεί τα καθήκοντά του όπως πρέπει στην ΕΚΤ, τότε υπάρχει μία διαδικασία δίωξης. Αλλά αυτό το αφήνω στις εθνικές αρχές και στην ΕΚΤ. Δεν είναι δικό μου θέμα. Το δεύτερο θέμα αφορά την καταπολέμηση του ξεπλήματος χρήματος. Υπάρχει ευρωπαϊκή νομοθεσία, πολύ καλή νομοθεσία, αλλά υπάρχει και ένα άλλο επιχείρημα για το ποιος είναι υπεύθυνος Είμαι υπέρ μιας ευρωπαϊκής αρχής που θα πρέπει να είναι υπεύθυνη για να μην υπάρχουν επιρροές εκεί που δεν πρέπει. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα μας ε, απασχολήσει. Υπάρχουν πολλές προτάσεις και αυτό φορά αυτούς που έχουν πολύ καλή γνώση για τις ροές χρήματος. Αυτές είναι οι κεντρικές τράπεζες, οι ευρωπαϊκή και οι εθνικές. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Ευχαριστώ πολύ. Ο Ραμόν Τρεμόσα. κύριε Κιόνι, καλώς ήρθατε. Άλλη μια φορά στο Κοινοβούλιο, έχω τρεις ερωτήσεις. Λοιπόν, πρώτη για τον Banco Popular. Πολλοί θεωρούν ότι κάποιοι κακοί υπολογισμοί στην έκθεση Deloitte του Ινού 17 ήταν ένας από τους λόγους για την εξηγένση του Banco Popular, της Banco Popular. Γιατί η Deloitte επελέγει εκ νέου για την έκθεση για το ότι κανείς πιστωτής δεν θα πρέπει να τα πάει χειρότερα. Δεύτερον, χρηματοδότηση κατά την εξηγένση υπάρχει ένα πρόβλημα χρονισμού. Γιατί χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να ληφθεί απόφαση για την εξυγέννηση και να γίνουν όλε οι αναγκαίε αποτιμήσει. Πώ θα μπορούσε να βελτιωθεί η χρηματοδότηση κατά την εξυγέννηση. Και τέλο, θέλω τη γνώμη σα για το εάν και κατά τόσο θα μπορούσε ο, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να ελέγχει τον ELA και όχι οι Εθνικές Τράπεζες. Ευχαριστώ. Τι καλά γερμανικά που μιλάτε, εγώ θα τολμούσα να σας απαντήσω ισπανικά. Λοιπόν, αυτοί οι κακοί υπολογισμοί για την έκθεση του επίπεδου 2, ναι, το αναγνώρισαν ορισμένοι, αλλά επειδή έχει ήδη απαντηθεί αυτή η ερώτηση. Είχαμε μια ανοιχτή διαφανή διαδικασία ανάθεσης επελέγει η Deloitte. Και δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ αποτίμησης 2 και αποτίμησης 3. Συντόμως θα δημοσιεύσουμε και την πρόσκληση προσφορών για την ε, αποτίμηση 3. Τώρα, πώς θα βελτιώσουμε την ε, χρηματοδότηση κατά την εξυγίανση. Ναι, πρέπει να το δούμε αυτό. Χρειαζόμαστε καλύτερα εργαλεία, ούτως ώστε σε περίπτωση εξυγένσης να διασφαλίζουμε ότι μετά την εξυγένση έχουμε επαρκή χρηματοδότηση. Αλλά νομίζω ότι αναφερθήκατε σε κάτι άλλο, στο οποίο θα είμαι πολύ προσεκτική. Αυτό το επιχείρημα ότι αν υπάρξει περισσότερος χρόνος μπορείτε να κάνετε καλύτερη εξολόγηση κτλ. Αλλά η περιπτώση εξυγίανσης αφορούν τράπεζες ε, που έχουν ε, λειτουργίες σε κρίσιμη κατάσταση που δεν ε, είναι δυνατόν να κλειδωθούν στον εαυτό τους για 4-6-8 εβδομάδες και μετά να πούνε να η λύση. Η χρηματοδότηση της εξυγέννησης είναι κάτι διαφορετικό. Πάντα, πάντα μου άρεσε αυτό το εργαλείο ε, παύσης, το λεγόμενο moratorium tool, για να κερδιθεί κάποιος χρόνος, τουλάχιστον δύο μέρες ας πούμε. Αυτό θα ήταν το σωστό εργαλείο αν δεν έχει ολοκληρωθεί η πώληση για παράδειγμα. Αλλά για την αποτίμηση δεν είναι το σωστό εργαλείο. Και όταν λέω προσωπικές απόψεις, ε, τελικά μετά το μετανιώνω. Αλλά δεν θα εκφραστώ για το αν ο ELA πρέπει να είναι ευρωπαϊκός ή εθνικός, δηλαδή να το διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ή οι εθνικές τράπεζες. Νομίζω ότι συνεργάζονται τους ή άλλους και μέχρι στιγμής τα έχουν πάει καλά. Ευχαριστώ πολύ. Έχω ένα λεπτό ακόμη. Στην περίπτωση της Banco Popular, εάν μπορούσατε να τα ξανακάνετε, τι θα είχατε κάνει διαφορετικά. Έχετε τίποτα από αυτού. Άψογη ερώτηση. Για ένα λεπτό. Η κυρία Κιόνιχ. Δεν θα είχα αλλάξει τίποτα. Ίσως για την ε, γνωστοποίηση θα είχαμε κινηθεί ταχύτερα, αλλά δεν θα αλλάξει τίποτα άλλο η απόφαση να απολυθεί η τράπεζα τη στιγμή που ελήφθη ούτω ώστε να διατηρηθούν και οι κρίσιμες λειτουργίες και η χρηματοπιστωτική σταθερότητα δεν θα είχαν κάνει τίποτα άλλο. Πάλι ένα ευρώ θα την είχατε πουλήσει, λέει ο κύριο Τρεμόσα. Θα την είχατε δώσει για ένα ευρώ στην Σανταντέρ. Είναι καλή τιμή. Κοιτάξτε, θα είμαι απόλυτα ουδέτερη. Ο καθορισμός της τιμής χρειάζεται έναν πολιτή που να είναι διατεθειμένος να ε, πληρώσει την τιμή. Και πάντα λέμε ότι ε, δεχόμαστε τον αγοραστή που προσφέρει την καλύτερη τιμή. Σβέν Γκίγκολτ. Σας ευχαριστήσω για την ε, αντισκεταστική αυτή ανταλλαγή απόψεων. Καταρχάς, να σας ευχαριστήσω για τα ξεκάθαρα σχόλια που κάνατε για την τοποθέτηση του Κοινοβουλίου σε σχέση και με την θέση του Συμβουλίου στο πακέτο για τις τράπεζες σε ό,τι αφορά τα δευτερεύοντα στοιχεία και και το grandfathering σε ό,τι αφορά τον έλεγχο των τραπεζικών κινδύνων τίθεται το θέμα αυτό. Σε ό,τι αφορά όμως το αποτέλεσμα που θα πετύχουμε στους τριμερείς διαλόγους, ανεξαρτήτως αυτού θα υπάρχει περιθώριο ελιγμού. Θα θέλαμε λοιπόν να γνωρίσουμε, να μας πείτε, θα μείνετε ε, άτεκτοι σε ό,τι αφορά το σεβασμό των προδιαγραφών από τις μεγάλες τράπεζες ε, Σε ό,τι αφορά την Τραπεζική Ένωση, θα ήθελα να μας πείτε κατά πόσο για τράπεζες που στο επιχειρηματικό τους μοντέλο περιλαμβάνουν μεγαλύτερο κίνδυνο σε ό,τι αφορά το οικονομικό έγκλημα και το ξέπλυμα βρωμικού χρήματος. Το λαμβάνετε αυτό υπόψη στις προτεραιότητές σας. Σε ό,τι αφορά την προετοιμασία της εξυγίανσης. Το λαμβάνετε αυτό υπόψη. Και τέλος γνωρίζουμε ότι στην παρούσα φάση και στο Eurogroup και στο, στην ΕΚΤ συζητούνται διάφορα ζητήματα σε ό,τι αφορά το πλαίσιο ρευστότητα για την εξυγίανση. Σύμφωνα και με το σχετικό πλαίσιο που είχε προταθεί. Είσαστε ενήμεροι για τι συζητήσει αυτέ και μπορείτε να μα ενημερώσετε ποιε είναι οι βασικέ λύσει που προτείνονται και ποιε είναι οι απόψει σα, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα επιμέρου στοιχεία μια ε, κοινή ε, ε, παροχή εγγυήσεων για ένα τέτοιο πλαίσιο ρευστότητα. Ευχαριστώ. Η απάντηση τη κυρία Κιόνι έχει να σας πω κατά πόσον θα παραμείνουμε αμετακίνητοι. Νομίζω ότι έχουμε πει εξ αρχή ότι το Emerald για μας είναι σημαντικό εργαλείο και ότι θα χρειαστούμε και από ποιοτική και από ποσοτική άποψη σωστή ποιότητα εργαλεία. Νομίζω ότι καταφέραμε να μετακινηθούν κάποιες τράπεζες και πολλές ε, τράπεζες ε, ε, προγραμματίστηκαν αντίστοιχα χωρίς να έχει ληφθεί η απόφαση. Άρα ναι, το ALM υπάρχει ως θέμα η EBRV νομίζω μας το επιβάλλει αυτό και στο SRV σε ό,τι αφορά τους κινδύνους που συνεπάγεται κάθε τράπεζα. Πρόκειται για μια τράπεζα η οποία βρίσκεται σε μια διαφορετική θέση σε ό,τι αφορά και το κεφάλαιο και την ρευστότητά της ή ενδεχομένω να μπει σε αυτή την κατάσταση. Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε το ενδεχόμενο να υπάρξουν τράπεζες με πολύ καλή κερδοφορία, αλλά με ένα επιχειρηματικό μοντέλο το οποίο ενδεχομένως να μην είναι επικίνδυνο, αλλά να ενέχει τον κίνδυνο γρήγορης πτώχευσης χωρίς έγκυρη προειδοποίηση. Αυτό λαμβάνεται λοιπόν υπόψη, αλλά πιστεύω ότι αυτό αποτελεί ένα θέμα για την επίβλεψη, προκειμένου να μην υπάρχει ένα τέτοιο υφέρπον στοιχείο, αλλά μπορεί να υπάρχει και μια ξαφνική τέτοια αλλαγή. Σε ό,τι αφορά το πλαίσιο ρευστότητα τη ESM, ξέρω ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εξετάζει το ενδεχόμενο αυτό, ότι γίνονται συζητήσει, αλλά εξ όσων γνωρίζω, ενδεχομένω φυσικά να έχω μείνει και λίγο πίσω, δεν έχει γίνει επίσημα τέτοια συζήτηση για το πλαίσιο ρευστότητας. Έχουν γίνει πολλές προπαρασκευαστικές εργασίες ακόμα συνεχίζονται. Είναι σαφές ότι όταν μιλάμε για τη χρηματοδότηση κατά την εξυγίανση, νομίζω ότι οι ίδιοι κανόνες που αναφέρθηκαν προηγουμένως για το μηχανισμό ασφάλειας ισχύουν. Θα πρέπει να είναι σαφές ότι αυτό χορηγείται στα πλαίσια της απόφασης εξυγίανσης με συγκεκριμένους όρους για να εξασφαλίσουμε ότι εφόσον ληφθεί η απόφαση εξυγίανσης, θα δίνουν τα χρήματα αυτά κατευθείαν. Πάντα αστευόμουν και έλεγα ότι ποτέ δεν θα δώσουμε χρήματα ε, το Σαββατοκυριακό χωρίς να ξέρουμε πώς θα έχει ρευστότητα την Δευτέρα. Είναι μια πολύ σημαντική συζήτηση η οποία όμως βρίσκεται σε μια πρώιμη φάση. Ευχαριστώ κύριος Βιέγκας. Τρία ερωτήματα έχω. Καταρχήν θα ήθελα να επανέλθω στις ελάχιστες απαιτήσεις για τους ίδιους πόρους και σε σχέση με το MRL, τις ελάχιστες απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων, θα ήθελα να ρωτήσω ποια είναι η διακριτική ευχέρεια του ΕΣΕ και πώς μπορεί να εφαρμόσει αυτές τις ελάχιστες, ελάχιστες απαιτήσεις που έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Σε σχέση τώρα με την διάρθρωση και τον συγκεντρωτισμό των τραπεζών, έχουμε ε, μία συγχώνευση μεταξύ ε, Unicredit της Ιταλίας και Societe Generale και αυτό μας ενδιαφέρει είναι να δούμε κατά πόσο αυξάνεται και ε, ο κίνδυνος ή πλέον έχουμε να κάνουμε με τράπεζες πολύ μεγάλες για να αποτύχουν. Δεν καταλαβαίνουμε γιατί, ε, γιατί προσφεύγουμε σε αυτές τις μεγάλες τράπεζες και δεν ξέρω κατά πόσο υπάρχουν άλλες δυνατότητες και ακαδημαϊκά ή τι πιστεύετε ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε για να παρέχουμε αυτές τις υπηρεσίες μέσα σε ίσως λίγο πιο διαφοροποιημένα πλαίσια. Ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Ως προς το ΕΜΡΕΛ δεν κατάλαβα ποια είναι η ερώτησή σας, αλλά θα πρέπει να υπάρχει η ευχέρεια να εντάξουμε το ΕΜΡΕΛ στην στρατηγική εξυγίανσης, αν είναι δηλαδή διάσωση με ίδια μέσα, αν είναι bail-in, μπορούμε να πούμε ότι θα γίνει επανακεφαλαιοποίηση της ε, τράπεζας για να υπάρξει αδειοδότηση. Γι' αυτό μιλάμε και για διπλές απαιτήσει κεφαλαιοποίησης και αυτό συμβαδίζει και με άλλα δικαιοδοτικά πλαίσια ως προς τις ε, στρατηγικές μεταφορών και πώληση τραπεζών, εδώ βρισκόμαστε σε πρόωρο στάδιο. Ως προς τη συγκέντρωση στον τραπεζικό τομέα, ε, δεν θα λάβετε απάντηση από μένα σε ενδεχόμενες φημολογίες, αλλά βλέπουμε ότι συρρυκνούνται οι τράπεζες. Βλέπουμε βλέως, βεβαίως συγκέντρωση τραπεζών που παρέχουν πολλές πιστοτικές ε, υπηρεσίες, οι οποίες βγαίνουν από την αγορά. Εμείς δεν ενθαρρύνουμε τη συγκέντρωση στην αγορά, αλλά οι αγορές κινούνται και τη στιγμή που δεν είναι ανησυχητική η κατάσταση, τότε δεν μας απασχολεί. Αλλά δεν σχολιάζω τη φημολογία. Και αυτή είναι μία από τις φήμες που ε, κυκλοφορούν. Σε σχέση με τις μεγάλες αυτές επιχειρήσεις, δούλεψα σε μία από αυτές 30 χρόνια πριν Και για να επανέλθω σε μια μεγάλη υπόθεση εξυγίανσης, είτε λάβετε την Banco Popular είτε οποιαδήποτε άλλη, τη στιγμή που χρειάζεται στήριξη, χρειάζεται η στήριξη πολλών ανθρώπων που δουλεύουν σε διάφορα δικαιοδοτικά όργανα, σε διάφορες χώρες. Άρα, το να μιλάμε για μικρότερες ε, επιχειρηματικές οντότητες, πολλές φορές δεν είναι δυνατή αυτή η προσφυγή. Υπάρχουν βεβαίως και πολλά δίκτυα όπου έχετε μεγάλες επιχειρήσεις στα κράτη-μέλη που συνεργάζονται εκ του σύνεγγης. Αλλά είναι μεγάλο το θέμα και δεν υπάρχει μία λύση. Μάρκο Βάλλη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Έχω τρία ερωτήματα προς την κυρία Κένιχ σε σχέση με το μηχανισμό ασφάλειας, το backstop αυτό θα πρέπει να δούμε τι μπορεί να γίνει, γιατί ακόμα και 60 δις δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν μία συστημική κρίση και ίσως θα έπρεπε να μας πείτε πώς θα έπρεπε να συγκροτηθεί ένα τέτοιο ταμείο εξυγίανσης. Πώς θα μπορούσαμε να έχουμε έναν αξιόπιστο μηχανισμό backstop. Δηλαδή, τι πρικοδοτήσεις θα πρέπει να έχει από την Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι ώστε να είναι αξιόπιστο αυτό το Ταμείο Εξυγίανσης όπως προς τη μείωση των κινδύνων επειδή δεν υπάρχει συγκεκριμένο ε, σχέδιο μείωσης κινδύνου που σχετίζεται με τίτλους ρευστότητας και ιδιαίτερα ως προς την φερεγγιότητα των τραπεζών, ιδιαίτερα της κεντρικής Ευρώπης και εδώ μιλώ για την μελέτη που έγινε για τη Γαλλία και τη Γερμανία, ο Ντράγκη μίλησε για τοξικά προϊόντα που εμπεριέχονται στα στοιχεία ενεργητικού των τραπεζών. Πιστεύετε λοιπόν ότι το backstop μπορεί να αντιμετωπίσει ένα τέτοιο συστημικό πρόβλημα. Και επίσης πώς έχουν οι ελάχιστες απαιτήσεις ΜΡΕΛ για τις ε, μεγάλες τράπεζες. Γιατί πρόκειται για τράπεζες που έχουν διαφορετικά εθνικά χαρακτηριστικά και ιδιαίτερα οι μικρές και ε, μεσαίες τράπεζες μεσαίας ε, κεφαλαιοποίησης κινούνται μεταξύ κεφαλαίων και καταθέσεων. Σας ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις ως προς το μηχανισμό ασφάλειας. Νομίζω ότι το μέγεθος του μηχανισμού στήριξης είτε είναι 60 είτε 70 ε, δις σε σχέση με το δικό μας ταμείο, το SRF, είναι κάτι που γίνεται ευρέως ε, κατανοητό για την κεφαλαιοποίηση. Ζούμε σε ένα διαφορετικό κόσμο από το 2008. Έχει αυξηθεί το κεφάλαιο των τραπεζών. Έχουμε το ε, MREL και ένα 8% δυνατότητα bail-in. Άρα υπάρχουν ρήτρες ασφαλείας πλέον. Και νομίζω ότι επαρκεί αυτή η δυνατότητα κεφαλαιοποίησης ή ανακεφαλαιοποίησης, αλλά αν χρειαζόσαστε τα χρήματα αυτά και τα χρησιμοποιήσετε για τη ρευστότητα, σε περίπτωση μεγάλων εθνικών τραπεζών θεωρώ ότι στην περίπτωση της ρευστότητας θα πρέπει να βρούμε μία άλλη λύση και εδώ μιλώ για τον δανειοδότη ίστα της καταφυγής, αν χρειαστεί. Δεν μπορώ να σας δώσω σαφείς αριθμούς. Τώρα, το δεύτερο ζήτημα, στο οποίο είχατε σταθεί και σε προγενέστερες ε, ε, συναντήσεις, ε, μιλάμε για στοιχεία ενεργητικού και ρευστοποίησή τους και εδώ θα πρέπει να δούμε πώς θα κινηθούν οι εποπτικές αρχές. Ε, πρόκειται για συγκεκριμένα ε, εγχειρήματα και μέσα που χρησιμοποίησε η ΕΚΤ που κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση. Στον προγραμματισμό εξυγίανσης έχει σημασία να δούμε κατά πόσο υπάρχουν τέτοια χαρτοφυλάκια και πώς πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Αλλά αυτό το θέμα μας απασχολεί εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα. Τώρα, πώς ορίζουμε το ΕΜΡΕΛ. Είναι ιδιαίτερα δαπανηρό για τράπεζες μεσαίας κεφαλαιοποίησης και θα ήθελα να πω ότι η πλειοψηφία των τραπεζών, για την πλειοψηφία των τραπεζών, η εξυγίανση δεν είναι η λύση, αλλά η διαδικασία εθνικής αφαιρεγγιότητας. Γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει αυτά τα μέτρα να εντάσσονται σε αυτό το πλαίσιο του ΕΜΡΕΛ και γι' αυτό δεν χρειάζεται επανακεφαλαιοποίηση αλλά διαδικασία αφαιρεγγιότητας. Για τις άλλες τράπεζες Λέμε ότι στις περισσότερες περιπτώσεις χρειάζεται επανακεφαλαιοποίηση, συμφωνείτε το πόσο και μετά βλέπουμε κατά πόσο το 25-26% προέρχεται από τα στοιχεία ενεργητικού και 12-13% από τις απαιτήσει κεφαλαίων. Αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε τις ε, στρατηγικές ε, μεταφοράς, αλλά όπως είπε και ο κύριος Τρεμόσα, δεν μπορούμε να βασιστούμε στην εξυγίανση με βάση το γνωμικό ότι θα προβούμε σε πώληση. Πάντα γίνεται πώληση στον καλύτερο αγοραστή, αλλά θα πρέπει να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε και τις καταθέσεις και ζητήματα που δεν απασχολούν τόσο πολύ τις μεγάλες τράπεζες. Μπαρμπαρα Κάπελ. Κυρία Κάνη, ε, καλή είναι η έκθεση για το 2017. Νομίζω ότι στην περίπτωση Banco Popular τα πήγατε πολύ καλά. Σωστά είπατε ότι η εξυγίανση έγινε έτσι που διατηρήθηκε η οικονομική σταθερότητα. Και αυτό δείχνει τη δυνατότητα δράσης του SRB. Το θέμα του Έμρελ πάντα μας ενδιαφέρει και το 17 και το 18 θα το παρακολουθήσουμε λοιπόν γιατί είναι σημαντικό. Και βεβαίως ε, και τα δευτερεύοντα MREL πρέπει να εξετάσουμε. Γιατί θέλουμε υψηλή ποιότητα και για τα MREL και για τους μηχανισμούς χρήσης τους. Και επανειλημμένα είπατε ότι οι τράπεζες οι ίδιες πρέπει να φροντίσουν ούτως ώστε να είναι εξηγιάνσιμες. Οπότε ερώτηση. Αν σας καταλαβαίνω καλά, προβλέπετε διπλασιασμό του SRB, SRF για τις δυνατότητες εξυγένσης. Δεν ξέρω, 60-70 δις προβλέπετε για το SRF μέσω των τραπεζών. Διπλασιασμός λοιπόν του SRF είτε μέσω πόρων είτε μέσω πιστοτικής γραμμής του ESM θα ήθελα να σας ρωτήσω, αυτός ο διπλασιασμός δεν τον επιλέξατε αυθαίρετα. Αυτά λοιπόν τα 60-70 δις σίγουρα κάπως τα βασίσατε σε υπολογισμούς. Μήπως θα μπορούσατε παρακαλώ να μας παρουσιάσετε την ανάλυση σας, ε, τους υπολογισμούς σας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Με συγχωρείτε γιατί ξεκίνησα να μιλάω γερμανικά. Ευχαριστώ για τα σχόλιά σας. Βεβαίως. Θα ε, μεταφέρω τα καλά σας λόγια για την έκθεσή μας στους συνεργάτες μου και χαίρομαι που κάποιος τη διάβασε. Για τα Emerald τώρα. Βεβαίως το θέμα της ε, ταξινόμησής τους μας απασχολεί. Θα είναι το θέμα που θα μας απασχολήσει, που μας απασχολεί ήδη για το 2018. Θέλουμε έναν ορισμό του ΕΜΡΕΛ για τα μεγαλύτερα πιστοτικά ιδρύματα εντός των πιστοτικών ομίλων. Είναι πολύ δύσκολο θέμα αυτό. Ε, Επικτηνόμεθα και σε ομίλους που δεν έχουμε ακόμη καλύψει και θα ε, έχουμε έναν ε, ορισμό ανά όμιλο. Είναι δύσκολο θέμα για το, το BRRD αυτή τη στιγμή δεν μας βοηθάει. Και το νέο πακέτο έχει κάποιους τομείς που δεν μπορούμε να γνωρίσουμε Τώρα για το διπλασιασμό του SRF. Υπάρχουν δύο θέματα. Δεν κάναμε κανένα τρομερό υπολογισμό. Βασιστήκαμε σε κάποια στοιχεία, τι χρειαστήκαμε κατά την προηγούμενη ε, οικονομική κρίση, τι ε, ε, ε επιπτώσεις θα είχε το 8%. Αλλά επίσης υπάρχει και μια πολύ λογική ε, παρατήρηση. Πρέπει να ξεπληρώσουμε ό,τι θα πάρουμε. Έτσι λοιπόν πρέπει να αισθανόμαστε άνατα ότι αν δανειστούμε από το ESM ή από οπωσδήποτε και αν ε, αποκαλείται όταν θα ε, μας δανείσει, θα πρέπει μεσοπρόθεσμα να το επιστρέψουμε. Δεν έχει καθοριστεί ακόμη Μπορεί να είναι τρία-πέντε χρόνια, αλλά δεν θα είναι μια αιωνιότητα. Πρέπει λοιπόν να μπορέσουμε να μοχλεύσουμε τον τραπεζικό κλάδο στο ποσοστό που μπορούμε να επιστρέψουμε. Είναι λοιπόν ένα backstop. Εάν δανειστείς, πόσα θα μπορέσεις μετά να συγκεντρώσεις χωρίς να μπει σε κάποιο φαύλο κύκλο. Άλλος ένας λόγος λοιπόν γιατί το backstop αυτό δεν μπορεί να είναι ε, απεριόριστου ύψου. Ευχαριστώ πολύ Ιάν Σαντέρ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ που έρχεστε τακτικά για να συζητήσετε μαζί μας. Δύο ερωτήσεις. Πρώτη. Η εκπόνηση σχεδίων εξυγένσης εργάζεστε από αυτού αυτή τη στιγμή για να, γίνει πιο, να γίνουν πιο λειτουργικά τα σχέδια εξυγίανσης των τραπεζών. Ξέρω ότι είναι πολλή δουλειά, ανάλυσης, επιλογής μέσων, στρατηγικών και θα πρέπει να γίνεται ουσιαστική εσωτερική εξυγίανση με αυτά που προτείνεται. Ποια είναι τα εμπόδια που αντιμετωπίζετε αυτή τη στιγμή στην εργασία σας και ποιες οι δυσχέρειες. Δεύτερη ερώτηση. Κυρία Πρόεδρε, συμφωνίες ε, συνεργασίας που ε, συνήψε το SRB με αμερικανικά και καναδικά συστήματα εγγύησης καταθέσεων. Μπορείτε να μας δώσετε περισσότερα στοιχεία για το περιεχόμενο αυτών των συμφωνιών και προβλέπετε να, να συνεργαστείτε και με άλλες δικαιοδοσίες. Και βεβαίως σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν έχουμε ένα έντις. Αυτό παρεμποδίζει την συνεργασία με άλλες περιοχές που έχουν παρόμοια συστήματα, που έχουν, τέτοια συστήματα. Λοιπόν, τα εμπόδια για την εξυγίανση. Ορισμένα τα έχουμε αντιμετωπίσει σε επιστολές που στείλαμε προς τράπεζες. Για παράδειγμα, πολλές φορές δεν έχουμε απλά πράγματα. Στη κάποια στοιχεία. Θέλουμε να μας στέλνουν οι τράπεζες μια φορά το χρόνο μια ε, λεπτομεριακή παρουσίαση των στοιχείων παθητικού. Αλλά όταν υπάρχει ενδεχόμενο εξυγένσης πρέπει να είναι αμέσως διαθέσιμα αυτά τα στοιχεία. Πρέπει λοιπόν να τα έχουν πάντα διαθέσιμα. Αυτό το αναγνωρίζουν όλες οι τράπεζες. Η, η υποδομή των ε, χρηματαγορών υπάρχουν τα clearing houses και όλες οι άλλες ε, όλες οι άλλες δυνατότητες. Είναι θέματα καθαρά ε, σωστής διαχείρισης και για τις πιο περίπλοκες, πιο μεγάλες τράπεζες, τουλάχιστον στο παρελθόν. Συχνά είχαν επιχειρηματικά μοντέλα και λογιστικά μοντέλα που αγνοούσαν την νομική πλευρά του θέματος. Θα πρέπει δηλαδή να μπορείς να διαχωρίσεις ε, τις ε, λειτουργίες σου. Είναι δουλειά εσωτερικής οργάνωσης και την αντιμετωπίζουμε. Συμφωνία συνεργασίας. Ε, βεβαίως. Έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία με το FTIC. Και τώρα πιστεύω ότι έχουμε το ίδιο επίπεδο συνεργασίας με το Federal Reserve Board, τους Καναδούς συναδέλφους. Και έχουμε μνημόνια συνεννόησης ή συνεργασίας και με άλλους. Αυτές οι συμφωνίες είναι όλες ε, μη δεσμευτικές, ε, τυποποιημένες διεθνείς συμφωνίες. Γιατί με βάση το καταστατικό μας πρέπει να το κάνουμε. Το χρειαζόμαστε αυτό για να ανταλλάσσουμε στοιχεία οι μεγαλύτερες τράπεζες ε, είναι τράπεζες που λειτουργούν σε διάφορες ε, δικαιοδοσίες. Πρέπει λοιπόν να μπορείς να ανταλλάξεις πληροφορίες. Αν εξετάσετε ε, τις συμφωνίες αυτές αναλυτικά θα δείτε ότι έχουν μια ρήτρα όλες αυτές. Ότι τα προσωπικά δεδομένα δεν συμπεριλαμβάνονται. Δεν τα χρειαζόμαστε για την συνήθεια εργασία μας αν τα χρειαστούμε για κάποιο λόγο, ε, απευθυνόμεθα στον ε, ε, επόπτη προσωπικών δεδομένων. Απλώς όμως ε, υπάρχουν κάποιες τυποποιημένες διατάξεις. Βεβαίως η συζήτησή τους και η σύναψή τους μας παίρνει πάντα πολύ χρόνο, αλλά είναι παρόμοιες. Και επεκτείνουμε αυτόν τον κατάλογο. Πρόσφατα υπέγραψα συμφωνίες με κάποιες μη ενωσιακέ τρίτες χώρες και συζητάμε και με κάποιες ασιατικές χώρες. Ο κατάλογος λοιπόν θα επιμηκυνθεί. Είμαστε σε λίγο διαφορετική κατάσταση από την ε, ΕΚΤΑΦ η οποία μπορεί να συμμετάσχει σε συμφωνίες που υπάρχουν στο εθνικό επίπεδο. Δεν υπήρχαν συμφωνίες για ε, αρχές εξυγένσης. Jakob von Weizsäcker. Ευχαριστώ, Πρόεδρε αξιότιμη κυρία Κιονέχια. Είναι τιμή μα και χαρά μα που είσαστε εδώ και ήταν και χαρά μα που διαβάσαμε την έκθεσή σα. Δύο ερωτήσει έχω να σα απευθύνω. Καταρχά, μια πιο γενική. Για τι στρατηγικέ ε, σκέψει ε, σε ό,τι αφορά την ε, φάση εξυγίανση και προφανώ. Από μία μεριά πρέπει να μπορούμε να, συνεργα... να συνεργαζόμεθα για να αποφευχθούν προβλήματα. Από την άλλη μεριά χρειαζόμαστε και μεγάλο βαθμό ε, έντονης ε, παρουσίας για να προστατευτούν οι επενδυτές όταν δεν λάμπει ο ιός, γιατί τώρα μεν λάμπει. Είναι λοιπόν ε, στοιχείο, είναι μια ε, πράξη εξισορρόπησης και θα ήθελα τη γνώμη σας για το κατά πόσο ε, είστε πιεστικοί έναντι, για παράδειγμα, των Ηνωμένων Πολιτειών. Συμφωνείτε ότι πρέπει, πρέπει να είστε. Ότι πρέπει να είμαστε αποφασιστικοί έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών. Και ότι είναι δύσκολο βέβαια σε αυτή την προσπάθεια επίτευξης ισορροπίας ίσως τελικά να μην είμαστε ιδιαίτερα αποφασιστικοί. Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση. Η δεύτερη ερώτηση λοιπόν τώρα σε ό,τι αφορά συγκεκριμένα το NCWO. Και αυτό παίζει σημαντικό ρόλο σε ό,τι αφορά και το Banco Popular, την τράπεζα. Όταν καταρτήσαμε και σκεφτόμασταν την εξυγίανση CCP, προσπαθήσαμε να καταβάλουμε μια προσπάθεια προκειμένου να λάβουμε υπόψη και τους συστημικούς, τις συστημικές επιπτώσεις σε ό,τι αφορά το NCWO με πιο λογικό τρόπο. Όταν εξετάζουμε λοιπόν το NCWO, την ε, αρχή αυτή, ότι κανένα πιστοτίζεται να μην βρίσκεται σε χειρότερη θέση, σε ό,τι αφορά τα τραπεζικά ζητήματα, τι διδαχτήκατε από την θέση του Κοινοβουλίου, την τοποθέτηση του Κοινοβουλίου σε ό,τι αφορά τα ζητήματα αυτά. Η απάντηση. Δεν είμαι βέβαιη κατά πόσο οι συναδελφοί μα, οι ομολογοί μα ε, στη ΣΥΠΑ ε, εστιάζονται πιο πολύ σε έναν τέτοιο κατάλογο αλλά έχουν διαφορετικό σύστημα. Ζητούν από τι τράπεζες να του αποδείξουν ότι είναι εξυγιάνσιμε υπό μια διαδικασία αφαιρεγκαιότητα. και εφαρμόζουν τα επιχειρήματα τα οποία προβάλλουν υπό τον τίτλο 2, υπό τη διευκόλυνση εξυγίανσης. Εγώ πιστεύω ότι λίγο πολύ ο νόμος μας η νομοθεσία μας βασίζεται στην ίδια αρχή. Είναι η τράπεζα εξηγιάνσιμη σύμφωνα με τη διαδικασία αφρικιότητας. Η JP Morgan, οι μεγάλες ε, τράπεζες της Αμερικής δεν ξέρω αν θα μπορούσαν να ακολουθήσουν μια τέτοια διαδικασία. Δεν το πιστεύω αυτό, αλλά αυτή είναι γενικώ η ιδέα και η αρχή. Εξετάζοντας λοιπόν τα διάφορα ζητήματα, διαπιστώνω ότι δεν είναι διαφορετική η προσέγγιση μας σε όλα αυτά τα θέματα. Θα είσαστε ενήμεροι ότι υπάρχει συνεργασία μεταξύ των Αμερικανικών αρχών της ε, Bank of England της Αγγλίας και ημών για να συζητήσουμε το πώς αντιμετωπίζουν διάφορα ζητήματα μεταξύ των οποίων και τον Μπέιλιν. Δεν έχω την αίσθηση ότι είμαστε σε διαφορετικό επίπεδο αντιμετώπισης. Εμείς βέβαια έχουμε μια πολύ πιο διαφοροποιημένη τραπεζική αγορά κοιτώντα την ε, Bank of England, το αμερικανικό σύστημα, για παράδειγμα, αυτοί επικεντρώνονται στην ε, ανώτερη βαθμίδα τραπεζών, όπου υπάρχει μεγαλύτερη ομοιογένεια, γιατί το FDIC καλύπτει την, ε, τη είπα και την τρατεντική ακτή, το σύστημα εγγύησης τραπεζών. Αυτή η αρχή που αναφέρατε. Για μας το θέμα αυτό μας απασχολεί ιδιαίτερως. Όταν ε, προβαίνουμε σε σχεδιασμό εξυγίανσης, ε, είναι σχεδόν αδύνατον, σχεδόν αδύνατον να δοθεί απόδειξη ότι δεν μπορεί να ληφθεί κάποια δράση για να μην βρεθεί σε χειρότερη θέση κάποιος πιστωτής. Γιατί στο σημείο αυτό τα πράγματα είναι διαφορετικά. Άρα το επιχείρημά μας ε, για την διοργάνωση των ελάχιστων απαιτήσεων δύο κεφαλαίων, το ένα MRL, είναι τα πιο φυσιολογικά κανονικά κριτήρια και κατά πόσον αυτό συνάδει με τα MRL. Δεν ήταν αυτό το σημείο κίνησης. Αλλά σήμερα επικεντρωνόμαστε κυρίως σε αυτό, σε αυτή τη μέθοδο. Αν υπάρχουν διάφορες δυνατότητες εξετάζουμε το ενδεχόμενο ανακεφαλαιοποίηση της τράπεζες, γιατί πολύ απλά και τα υπόλοιπα εργαλεία προαπαιτούν άλλες διεργασίες. Τώρα, για να είμαι ειλικρινής, ε, δεν ξέρω να σας απαντήσω και θα πρέπει να ξαναεξετάξω το έγγραφο της εξυγίανσης CCP για να το χρησιμοποιήσουμε στους περαιτέρω συζητήσει Μια και βρισκόμαστε στην διαδικασία του τρομερού διαλόγου, θα σα ενημερώσω κατά πόσο υπάρχει κάποια συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ, κύριο Κάρα. Προέντρε, κυρία Κιόνιγκ. Είναι πράγμα ευχάριστο και καθησυχαστικό να σας ακούμε γιατί είσαστε πάρα πολύ αντικειμενικοί στην απάντηση των ερωτήσεων. Έχω δύο συμπληρωματικέ ερωτήσει να κάνω. Καταρχά, ό,τι αφορά την αφαιρεγκαιότητα και κατά δεύτερον, μια ερώτηση για την ανταλλαγή πληροφοριών. Καλώ ορίζετε την ανάγκη να υπάρχει ένα ενιαίο δίκαιο, μια ενιαία νομοθεσία για την αφαιρεγκαιότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι το τέλος ε, το 2018 θα πρέπει να υποβάλει σχετικές προτάσεις. Αλλά πείτε μας εσείς ε, από την πολιτική ηγεσία τι θα επιθυμούσατε. Γιατί δεν θεωρείτε ότι χρειαζόμαστε και γενικά μια εναρμόνιση του σχετικού δικαίου μεταξύ των κρατών. Κατά δεύτερον, για την ανταλλαγή πληροφοριών. Είσαστε στη φάση επεξεργασίας αυτού του μνημονίου συμφωνίας ε, κατανόησης μεταξύ ΕΚΤ για τη βελτιωμένη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εθνικών αρχών εξυγίανσης. Τι πιστεύετε? Αυτό το Memorandum of Understanding μέχρι πότε πιστεύετε θα ολοκληρωθεί? Again. Σας ευχαριστώ. Θα απαντήσω στα αγγλικά. Δύσκολο. Δύσκολο να ακούμε τη μητρική μας και μετά να μιλήσουμε σε άλλη γλώσσα. Για την αφαιρεγγιότητα. Το ξεκαθαρίσαμε, πιστεύω. Χρειάζεται κατεπηγόντως εναρμόνιση και μαζί με αυτήν κάποιες βέλτιστες πρακτικές για την διαδικασία αφαιρεγγιότητα στις τράπεζες. Το λέω αυτό όμως πάντα και πιστεύω ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ ρεαλιστές ότι αυτό δεν εμποδίζει τα κράτη-μέλη να επιλύσουν οποιαδήποτε θέμα τα πιστεύουν θα πρέπει να επιλύσουν και στη εθνική νομοθεσία για την αφαιρεγγιότητα και στις εθνικές διεργασίες που προβλέπονται. Τώρα, για να μιλάμε για να μιλήσουμε για καθεστώς αφαιρεγγιότητας για χώρες. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον μεν, αλλά θα ήμουν πολύ ικανοποιημένη αν μέχρι τα τέλη του 2018 είχαμε μια διαδικασία εξυγίανσης για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και ούτε καν για όλα. Έχω λοιπόν την προσωπική μου άποψη για τα θέματα αυτά, για την ανταλλαγή απόψεων και πληροφοριών συγγνώμη, μεταξύ του ενιαίου Συμβουλίου Εξυγένσης και της ΕΚΤ. Έχουμε δημοσιεύσει την αναθεωρημένη αυτή η συμφωνία μεταξύ ΕΚΤ και Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανση. Το θετικό στοιχείο είναι ότι η συνεργασία αυτή έχει προχωρήσει τα τελευταία τρία χρόνια και έχουμε λάβει υπόψη ε, ουσιαστικά ένα πράγμα το οποίο καταδεικνύει ότι τα πράγματα κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση. Έχουμε πλέον πολύ μεγάλο όγκο αυτοματοποιημένων πληροφοριών που ανταλλάσσονται. Δεν χρειάζεται καν να προβούμε σε σχετικό αίτημα Φυσικά υπάρχουν ε, πολλά θέματα ακόμα στα οποία χρειάζεται να στείλουμε ένα αίτημα για την παροχή πληροφοριών, αλλά δεν χρειάζεται και τεκμηρίωση. Απλά αναφέρουμε ποιε πληροφορίε χρειαζόμαστε. Και αυτέ οι πληροφορίε, για να είμαστε ακριβεί, είναι πληροφορίε συμπεριλαμβάνοντα τα δεδομένα εποπτείας, ε, δεδομένα SSM, τα οποία είναι τμήμα των δεδομένων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αλλά από πλευράς δικιάς μας ε, χρειάζεται να προβούμε σε έτοιμα για την παροχή των πληροφοριών αυτών. Τα πράγματα πηγαίνουν πάντα καλά. Εξακολουθώ, ωστόσο, να τονίζω ότι μας προσκαλούν και σε πολλές ε, συνεδριάσεις ε, SSM και εξακολουθώ να πιστεύω ότι χρειάζεται αμοιβαιότητα. Και εμείς δηλαδή να είμαστε μόνιμοι παρατηρητές των συνεδριάσεών τους, όπως και αυτοί είναι μέλη και μόνιμα, μόνιμοι μόνιμα παρακολουθούν τις δικές μας συνεδριάσεις. Αυτό θεωρώ ότι είναι καλό επιχείρημα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σφρουντσούλητσα. Ε, Σας ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, χαίρομαι γιατί βλέπω ότι η ε, αποστολή του ΕΣΕ σχετίζεται με την εξυγίανση του τομέα των δημοσίων οικονομικών και εντάσσεται στα πλαίσια της Τραπεζικής Ένωσης. Θα ήθελα να πω ότι έχουμε πολύ δρόμο να διανύσουμε για την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης με βάση το έγγραφο του Ιουνίου του 2016. Θα πρέπει να θέσουμε σε εφαρμογή το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εγγύησης των Καταθέσεων και θα πρέπει να σας πω ότι αυτή είναι η στιγμή για να συνεχίσουμε να ασκούμε πίεση για την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εγγύησεων των Καταθέσεων θα πρέπει να οδηγήσει στην πλήρη χρηματοδότηση της ρευστότητας και αντιστάθμιση των ε, κινδύνων καθώς και των απολειών. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία για να έχουμε σωστή και αποτελεσματική λειτουργία της ε, εποπτείας και της εξυγίανσης είναι η εκτουσίνεγκης παρακολούθηση του συστήματος. Επίσης, χρειάζεται ένας μηχανισμός ασφάλειας που ορίζει το ενίο Συμβούλιο Εξυγίεσης. Πράγματι, κυρία Πρόεδρε, οι τράπεζες ξέρουν πολύ καλά τι πρέπει να γίνει για να εξυγιανθούν. Και χαίρομαι διότι οι ομάδες διαχείρισης εργάζονται σε αυτό τον τομέα. Τη στιγμή που η συμμετοχή των τραπεζών ε, έχει μεγάλη σημασία, ποιες είναι οι δράσεις που προβλέπονται στην επόμενη περίοδο, έτσι ώστε να υπάρχει στενή συνεργασία στον τομέα αυτό. Απάντηση. Θα προσπαθήσω να σας απαντήσω. Δεν υπάρχει καμία διαφωνία ως προς το ότι δεν υπάρχει ακόμα ο τρίτος πυλώνας της Τραπεζικής Ένωσης. Θα πρέπει να γίνει πραγματικότητα και δυστυχώς δεν υπήρξε και μεγάλη κινητικότητα το 2017-18 μέχρι τώρα. Ας ελπίσουμε λοιπόν να συνεχιστεί αυτή η διαδικασία για το σωστό backstop. Το συζητήσαμε και έχουμε ταχθεί υπέρ της επίλυσης του ζητήματος. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για μηχανισμό ασφάλειας του ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης στο τέλος της διαδικασίας αμοιβαιοποίησης. Όχι τώρα δηλαδή, αλλά για το τέλος αυτής της φάσης, η οποία θα επιταχυνθεί. Και τέλος, όπως είπατε πολύ σωστά, οι τράπεζες γνωρίζουν πολύ καλά, χάρη και στις ομάδες μας, που καθιστούμε σαφές στις τράπεζες τι πρέπει να κάνουν και, ξέρει, και ξέρουν οι υπεύθυνοι τι πρέπει να κάνουν μέσα στα πλαίσια μίας ε, σωστής διαχείρισης. Θα πρέπει λοιπόν να ε, ασχοληθούν με συγκεκριμένα θέματα και μετά να ορίσουν ένα χρονοδιάγραμμα επίλυσης. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος. Δεν μπορείτε να αποστείλετε μία επιστολή που να λέτε σε μία τράπεζα «Μα εγώ ξέρω καλύτερα πώς να εξηγιανθείτε» και θα το κάνετε με αυτόν τον τρόπο. Αυτό θα γίνει μόνο με ε, διάδραση και εποπτεία. Ζητώ συγγνώμη για αυτό το θόρυβο. Ε, χαίρομαι για το, για το t-shirt που βλέπω του συναδέλφου Μανέτιτς. Ίσως οι Βρετανοί να μην το εκτιμούν ιδιαίτερα. Αλλά σας παρακαλώ πολύ να μην κάνετε ε, θόρυβο. Brian Hayes. Χαιρόμαστε που σας βλέπουμε πάλι. Μία ερώτηση σε σχέση με το MREL και το Brexit. Ξέρω ότι δεν μπορείτε να πείτε πολλά, αλλά υπάρχει μεγάλη ε, ανησυχία. Η, τα στοιχεία παθητικού ίσως να μην μπορέσουν να αντισταθμιστούν μέσω ΕΜΡΕΛ. Άρα ίσως υπάρχει ε, μη διασφάλιση με βάση το ΕΜΡΕΛ μετά το Brexit πολλές ε, ε, τράπεζες και στην Ιρλανδία, στη χώρα μου, αλλά και σε ολόκληρη την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν πολλά στοιχεία παθητικού δυνάμει του ευρωπαϊκού δικαίου και θα θέλαμε να μας πείτε κατά πόσο το Συμβούλιο Εξυγίανσης μπορεί να μας δώσει εγγυήσεις επί του θέματος γιατί η τράπεζες θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στις διεθνείς αγορές και μετά το Brexit. Χρειάζεται ε, βεβαίως ή ίσως μία διασφάλιση μέσω νομοθεσίας έτσι ώστε να λάβουμε υπόψη τι ισχύει σε περίπτωση των οφειλών δυνάμει του Βρετανικού δικαίου. Σε μία τέτοια περίπτωση ίσως θα πρέπει να προωθήσουμε το ε, grandfathering. Αλλά θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε τι θα γίνει με τα στοιχεία παθητικού. Απάντηση. Πολύ σκόπιμη η ερώτηση και φυσικά είναι ερώτηση επί της ουσίας ως προς το Brexit. Αυτή τη στιγμή έχει αρχίσει ο διάλογος με τις τράπεζες έτσι ώστε να ε, δούμε ποια είναι τα στοιχεία παθητικού και τι ομολογίες έχουν εκδοθεί. Μας διέπει το βρετανικό δίκαιο στη συγκεκριμένη περίπτωση και όπως είπατε πολύ σωστά, η καλύτερη λύση θα ήταν καθαρά νομική υφής, το grandfathering, που αναγνωρίζει τις αποφάσεις εξυγίανσης κατά τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Διαφορετικά, αν θεωρήσουμε ότι θα έχουμε ένα σκληρό Brexit, τότε από την ημέρα του Brexit τα ζητήματα αυτά ε, δεν θα υπάγονται στο δικό μας MREL, γιατί δεν θα μπορέσει να τεθεί σε εφαρμογή. Βεβαίως, για τις νέες εκδόσεις ομολογιών, και αυτό το είπαμε στις τράπεζες πέρσι, για τις νέες εκδόσεις, εάν δεν υπάρχει νομική ασφάλεια, τότε θα πρέπει να θεωρήσετε ότι υπάρχει μια συμβατική ρήτρα. Το δύσκολο είναι οι ομολογίες που προϋπάρχουν είναι εύκολο να πείτε θα προσθέσω μία ρήτρα, αλλά δεν είναι κάτι το εύκολο. Και η θέση μας είναι ότι εποπτεύουμε την κατάσταση, προειδοποιούμε τις ε, τράπεζες γνωρίζοντας ότι μερικές μικρές τράπεζες δεν γνωρίζουν καν την ύπαρξη του προβλήματος και επίσης το βλέπουμε και εσωτερικά. Να δούμε δηλαδή πώς ορίζονται αυτές οι λήξη πρόθεσμες ομολογίες, πότε λήγουν δηλαδή. Εν πάση περιπτώσει θα υπάρχει μια μεταβατική φάση και πιστεύω και ευφυείς νομικές ε, λύσεις. Και βεβαίως ε, απευθύνω το θέμα και σε εσά. Ευχαριστώ. Τελευταία ερώτηση και σχόλιο. Πολύ λογικά αυτά που είπατε για την ε, σύνδεση της εξυγίανσης με τα άλλα θέματα που είναι ε, διαφορετική από την ανακεφαλαίωση, ανακεφαλαιοποίηση. Έχουμε το 8% και συμφωνώ απόλυτα με εσάς ότι η αξιοπιστία ενός μηχανισμού ασφαλείας, ενός backstop εξαρτάται από το θα είναι από το κατά πόσο θα είναι διαθέσιμο. Αλλά αυτό είναι μια εξάντια αιρεσιμότητα. Εσείς θα την ε, αξιολογήσετε. Όχι εσείς. Όχι κάποιος άλλος. Οπότε είναι πολύ περίπλοκο να έχουμε ένα αποτελεσματικό τέτοιο μηχανισμό backstop. Επίσης, ενδιαφέρον αυτό που είπατε, ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε το θέμα της χρηματοδότησης τη εξυγίανσης. Μπορείτε να μας πείτε κάτι περισσότερο για αυτά, αλλά και κάτι άλλο, που είναι η χρηματοδότηση για να αποφευχθεί η εξυγίανση. Ε, γιατί το ξεχνάμε λιγάκι. Έχουμε τον ELA, ε αλλά έχουμε και το άρθρο 32 που μπορεί να μας δώσει χρηματοδότηση. γιατί φοβάμαι ότι έχουν χάσει κάθε περιεχόμενο αυτές οι δυνατότητες, γιατί μπορούν να μας βοηθήσουν να αντιμετωπίσουμε ένα μεγαλύτερο πρόβλημα χρηματοδότηση τη ίδια εξυγίανση. Ευχαριστώ για τα ενθαρρυντικά σας λόγια, για την ε, αξιοπιστία του backstop. Θα ε, το επαναλάβω παντού και ελπίζω να γίνει κατανοητό. Η χρηματοδότηση της εξυγίανσης είναι, όπως ήδη είπα, ένα θέμα που μόλις άρχισε να συζητιέται. Είναι θετικό ότι η Κεντρική Τράπεζα σκέφτεται να υπάρχει μια διευκόλυνση για την χρηματοδότηση της εξυγίανσης. Αλλά αυτό το θέμα θα πρέπει να μας απασχολήσει και πριν από την εξυγένση και κατά την εξυγένση. Όπως είδαμε στο παρελθόν. η χρηματοδότηση της προεξηγένσης αν συνεχιστεί μπορεί να καταστήσει πιο ε, δαπανηρή και πιο περίπλοκη την εξυγίανση την ίδια. Δηλαδή, πρέπει να διαλέξουμε καλά το σημείο πότε θα ληφθεί η απόφαση για να ξεκινήσει η εξυγίανση. Χρειάζεται η εξυγίανση δηλαδή ή μπορεί να διατηρηθεί ε, μια τράπεζα ως έχει ε, αναμένοντας μια ιδιωτική λύση. Νομίζω ότι μια προβληματική τράπεζα δεν βοηθιέται πάντα αν περάσει εξυγίανση. Ε, μπορεί να είναι αποτρεπτικό μιας πρώτερης λύσης. Πρόεδρος, ναι, το θέμα είναι εάν ε, το πρόβλημα χρηματοδότησης είναι απλώς κάτι παροδικό ή αν σχετίζεται με την φερεγγιότητα της τράπεζας. Αλλά χαίρομαι που συμφωνείτε ότι υπάρχουν και δύο διαστάσεις. Και φυσικά η προεξηγιανική χρηματοδότηση είναι περίπλοκη και αυτή. Γιατί πρέπει να διακρίνει κανείς ε, μεταξύ των δύο κατηγοριών. Αλλά υπάρχει το πρόβλημα. Και είναι θετικό ότι τουλάχιστον αναγνωρίζεται και ότι συζητιέται. Σας ευχαριστώ πολύ. Πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση η οποία λύγει εδώ και σας ευχόμαστε καλές διακοπές και να διακόψουμε για δύο λεπτά πριν ξεκινήσουμε την ψηφοφορία.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 αγαπητοί συνάδελφοι. Πολύ ωραία εικόνα. So, uh, Αγαπητοί συνάδελφοι, περνάμε στι ψηφοφορίε. Θα κάνουμε μια δοκιμαστική ψηφοφορία καταρχήν. Δοκιμαστική άρχεται. Ορισμένοι συνάδελφοι ακόμη δεν έχουν ψηφίσει. Ψηφίσατε όλοι παρακαλώ. Ψηφίστε παρακαλώ τουλάχιστον για τη δοκιμαστική, όσοι έχετε την κάρτα σας. Λείπουν δύο. Α, έχουν ε, βάλει στο μηχάνημα την κάρτα τους, αλλά δεν έχουν ψηφίσει. Σας παρακαλώ ψηφίστε για να δούμε τους παρόντες από πλευράς ομάδων. Σας παρακαλώ ψηφίστε. Ωραία. Λοιπόν, πέρασε. Ωραία. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Πρώτο θέμα, η αναδιαβούλευση για την επιτυχή ολοκλήρωση του τριμερούς διαλόγου για θέματα ανταγωνισμού. ECN Η Εισηγητής είναι ο Ανδρέας Σουάμπ. Θα ήθελε να πει κάτι. Παρακαλώ, Ανδρέας, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εσά και όλου του συναδέλφου που με βοηθήσατε. Ήταν πολύ επικοδομητικό ο τριμερή διάλογο με το Συμβούλιο. Νομίζω ότι επιτύχαμε έναν καλό συμβασμό, συνολικά ισορροπημένο, περισσότερη εξαρτησία για τι αρχέ ανταγωνισμού, ανταγωνισμού τι εθνικέ περισσότερους ανθρώπινους πόρους και πόρου και ενισχύουμε την πολιτική ανταγωνισμού συνολικά. Επί ενό σημείου θέλω να επιστήσω την προσοχή σα τα ενδιάμεσα μέτρα. Γίνεται μια συζήτηση ιδιαίτερα στα πλαίσια της ψηφιακής οικονομίας και πώς θα βοηθούσαν την Επιτροπή να δρά ταχύτερα. Επιτύχαμε ότι θα υπάρξει μια δήλωση της Κομισιόν στο Κοινοβούλιο για το θέμα αυτό. Είναι τμήμα της συμφωνίας και αυτό μας ικανοποιεί ιδιαίτερα και με πολύ χαρά το προτείνω ε, για να το υπερψηφίσετε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, λέει ο κύριε Σιγητά και συγχαρητήρια. Ήταν πολύ θετική η κατάληξη. Έχουμε το κείμενο της δήλωσης της Επιτροπής εδώ. Για να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα. Δεν θα το διαβάσω. Νομίζω ότι είναι πολύ θετική η κατάληξη. Να ψηφίσουμε λοιπόν το συμφωνηθέν κείμενο. Στα πλαίσια των διοργανικών διαπραγματεύσεων, ονομαστική ψηφοφορία άρχεται. Πέρας. 44 υπέρ, 4 κατά. Και δεν είδα τις αποχές. Εντάξει όμως ε, καταγράφει και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Θα δούμε λοιπόν και πόσες αποχές. 44 υπέρ, 4 κατά και 4 αποχές. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Τώρα να περάσουμε στην έκθεση του Φαντελ Κέντελαρ για το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας όσον αφορά τα ειδικά καθεστώτα για τις μικρές επιχειρήσεις. Τροπολογία 4 υπέρ παρακαλώ. Κατά. Είστε υπέρ μάλιστα. Ωραία. Ελέγχουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 33 υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 5 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 35 υπέρ κατά αποχές δεν βλέπω τι κάνει το ΕΛΚ. Καλά, να ελέγξουμε. Ελέγχουμε την 35. Νομίζω ότι θα εγκριθεί τότε, αλλά... Πέρας. Απορρίπτεται. 34. Υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 36. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 37. Υπέρ. Κατά Αποχές. Απορρίπτεται. Να ελέγξουμε. Καλά. Ελέγχουμε την 37. Πέρας. Απορρίπτεται. 6. Υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. 39 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 40 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 41 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 42 υπέρ κατά αποχές α όχι ελέγχουμε τη 42 πέρας εγκρίνεται 44 υπέρ κατά ελέγχουμε τη 44 Πέρας. Εγκρίνεται. Οπότε περάμε 46 υπέρ, κατά αποχές, απορρίπτεται. 47 υπέρ, κατά ελέγχουμε 47. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 48 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική α υπέρ κατά συμβαστική α εδώ λέει μείον στηρίζεται μόνο από δύο ομάδες ελέγχουμε τη συμβαστική α άρχεται πέρας εγκρίνεται 50... Ε, α, όχι. Α, συγγνώμη, δεν ε, το αναφέρω κατάλληλο ψηφοφοριών. Περνάμε στην 52. Υπέρ, κατά, ελέγχουμε. Την 52. Πέρας. Δεκτή. 10 υπέρ κατά αποχές δεκτή 54 υπέρ κατά ελέγχουμε την 55 πέρας δεκτή 12 υπέρ κατά αποχές δεκτή 58, 59 και 13 υπέρ κατά αποχές δεκτές. 60 και 14 υπέρ κατά αποχές δεκτές. 15 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 16 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 17 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 18 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 19 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 20 υπέρ κατά απο... Ελέγχουμε την 20. Πέρας. Δεκτή. 21 υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται. 22 υπέρ κατά αποχές. Δεκτή. 23 υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται. 24 υπέρ κατά Πράσινα κατά. Καλώς, ελέγχουμε. Την 24. Πέρας. Απορρίπτεται. Δύο ψήφοι διαφορά. 25 υπέρ κατά αποχές. Δεκτή. 26 υπέρ κατά αποχές. Δεκτή. 3 υπέρ κατά αποχές. Δεκτή. Περνάμε στην 30 υπέρ. Κατά ελέγχουμε. Την 30. Άρχεται. Πέρας. Ισοψηφία απορρίπτεται. 31. Υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Ψηφίζουμε την τροποποιηθήσα πρόταση της Επιτροπής, ονομαστική άρχεται. Πέρας. 44 <coughs> υπέρ, 4 κατά 4 αποχές. Συγχαίρουμε τον εισηγητή. Και τώρα να περάσουμε στο σχέδιο έκθεση ε, του Brian Hayes για τη σχέση μεταξύ τη Ευρωπαϊκή Ένωση και των τρίτων χωρών σχετικά με τη ρύθμιση και την εποπτεία των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Συμβαστική Α. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική Β υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική Σ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 60 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 61 ε, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 62 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 63 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Αρχικό κείμενο. Υπό παράγραφος 2, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική D, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική F, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμ... Τροπολογία 78, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική G, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική H, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 89 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 91 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική για τα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική J υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική K υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 119 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται. Συμβαστική L υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική μη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική νη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική όμικρον υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική πι ρο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική Q υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 162 υπέρ κατά Έλεγχος παρακαλώ για την 162. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική R. Υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 172 υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. Απορρίπτεται, συγγνώμη. Συμβαστική S υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. Συμβαστική T τάφ υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. Συμβαστική U υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. Τροπολογία 194 υπέρ κατά. Έλεγχος παρακαλώ για την 194. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Πέρασε απορρίπτεται. Συμβαστική Β, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 200. CP2. Προφορική τροπολογία. 200 ε, παρακαλώ, υπέρ, κατά αποχές, απορρίπτεται. 206 υπέρ, κατά αποχές, απορρίπτεται. 207 υπέρ, κατά αποχές, Έλεγχος παρακαλώ για την 207. Πέρας. Απορρίπτεται με μία ψήφο διαφορά. 208 υπέρ. Κατά. Το ΕΛΚ τι ψηφίζει, εγκρίνεται. Σεμιβαστική W υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 212 υπέρ κατά. Υπέρ για τη 212 κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Έλεγχος παρακαλώ για την 212. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Α, είσαστε υπέρ. Γιατί είδα το πλήν. Πέρασε. Απορρίπτεται. Σε χ, υπέρ, κατά, αποχές, έγκρινεται. 220, υπέρ, Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική υψηλών υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 230 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 231 υπέρ κατά. Έλεγχος παρακαλώ για την 231. Πέρας. Απορρίπτεται. Αρχικό κείμενο, παράγραφος 24. Ψηφίζουμε υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 1 έως 8 αιτιολογική σκέψη υπέρ. Κατά. Έλεγχος. Ετυλογικές σκέψεις 1 έως 8. Α, δικό μου λάθος, λέει ο πρόεδρος. Νόμιζα ότι ήσασταν κατά. Πέρας ψηφοφορία. Εγκρίνεται φυσικά. Χωρί μεγάλη διαφωνία. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Έλεγχος παρακαλώ για την τροπολογία υπερθμών 3. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική Ζ, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική αλφα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 10, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική β, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική AC, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 16, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Απορρίπτεται, συγγνώμη. Τροπολογία 18 υπέρ κατά απόχέ. απορρίπτεται. Συμβαστική ΑΔ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 23 υπέρ κατά Έλεγχο παρακαλώ για την 23. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται τροπολογία 25 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έγκρινεται 26 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 27 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 28 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος παρακαλώ για την 28. Ψηφίζουμε. Πέρας. απορρίπτονται. ΑΕ, συμβαστική υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 33 υπέρ, κατά αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 34 υπέρ, κατά. Έλεγχος παρακαλώ. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για την 34. Πέρας. Απορρίπτεται Τροπολογία αρχικού κειμένου, ε, λογική σκέψη G, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 38, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τώρα, το σύνολο του κειμένου, όπως τροποποιήθηκε, με ονομαστική κλίση. Ψηφίζουμε, παρακαλώ. Πέρας. 46 ψήφοι υπέρ, 4 κατά, 2 αποχές. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Και έτσι ολοκληρώσαμε τις ψηφοφορίες. Να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα μέχρι τις 5 και 5 τέταρτο, όπου θα έχουμε και μαζί μας ε, τους ε, την, τον Υπουργό της Αυστρίας. Διάλειμμα λοιπόν 45 λεπτών.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

Dear colleagues. Αγαπητοί συνάδελφοι, καλώς θερμά τον ε, Αυστριακό Υπουργό Οικονομικών Χάρτζη Κλόγκα, που όπως ξέρετε είναι και πρόεδρος ε, του Συμβουλίου ΕΚΟΦΗΝ για το τρέχον εξάμεινο. Ευχαριστώ που δεχτήκατε την πρόσκλησή μας να παρουσιάσετε τις προτεραιότητες της ε, Αυστριακής Προεδρίας στους τομείς ε, ενδιαφέροντος της ΕΚΟΝ που είναι πολύ ευρύ, ευρύς και καλύπτουν ε, πολλά βασικά θέματα που μας απασχολούν και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Eurogroup και το ECOFIN φυσικά όλους. Χαίρομαι που έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε αυτή την ανταλλαγή απόψεων που θα καλύψει φυσικά γενικότερα τις προτεραιότητές σας, αλλά σίγουρα θα εστιάσει στους τριμερείς διαλόγους που είναι η τελευταία φάση της διαδικασίας συναπόφασης για το τραπεζικό πακέτο. Οπότε έχετε ιδιαίτερα απαιτητικά καθήκοντα ως Προεδρία γιατί επειδή πλησιάζουμε στην λήξη της θητείας ε, έχουν συσσωρευτεί πολλά νομοθετικά θέματα και δεν είναι μόνο θέμα ποσότητας αλλά και ποιοτικά είναι πολύ σημαντικά οπότε εκτιμούμε ιδιαίτερα τον πολύ θετικό και ανοιχτό τρόπο με τον οποίο η Προεδρία σας αντιμετωπίζει τα θέματα αυτά και το διάλογο με το Κοινοβούλιο Διαβάζοντα τα πορίσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ωστόσο, δεν μας ε, ικανοποίησε τόσο πολύ η διατύπωση ότι η γενική προσέγγιση του Συμβουλίου είναι πιο σημαντική από τη στάση του Κοινοβουλίου. Νομίζω ότι είμαστε δύο συνομοθέτες. Ε, οι ΜΕΝ εκπροσωπούμε απευθείας τους ε, Ευρωπαίους πολίτες και οι άλλοι τα κράτη-μέλη. Είμαστε ισότιμοι Συνομοθέτε. Εκτιμώ λοιπόν που η Προεδρία σας εκκινεί με ανοιχτό και επικοδομητικό τρόπο την συζήτηση αυτή. Τουλάχιστον ε, αυτή είναι η αρχική σας προσέγγιση γιατί η συζήτηση μόλις τώρα έχει ξεκινήσει. Εκτιμώ ιδιαίτερα τη θετική σας προσέγγιση. Έχουμε το τραπεζικό πακέτο, αλλά και η Ένωση Κεφαλαίου Αγορών είναι πολύ σημαντική, το InvestEU πολλά ε, κρίσιμα νομοθετικά θέματα. Σας εύχομαι λοιπόν κάθε επιτυχία για αυτά τα τόσο απαιτητικά καθήκοντα που έχετε εντοπιό σας και για τον ε, ρόλο διεύθυνσης ε, των συζητήσεων στο Συμβούλιο και εμείς ως Κοινοβούλιο θα επιδιώξουμε να είμαστε επικοδομητικοί, ρεαλιστικοί και έτοιμοι να δεχθούμε συμβιβασμούς γιατί η Ευρώπη χρειάζεται αποφάσεις. Χρειάζεται να καταλήξουν μια σειρά από θέματα, ένα καλύτερο πλαίσιο τραπεζικής ένωσης, ένα ενιαίο εγχειρίδιο κανόνων για τις κεφαλαιαγορές, για να έχουμε περισσότερες επενδύσεις. Είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξο γιατί πιστεύω ότι θα συνεργαστούμε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ και σας δίνω το λόγο για την εισαγωγική σας ε, ομιλία. Κύριε Πρόεδρε μου. κύριοι βουλευτές, κυρίες και κύριοι βουλευτές, χαίρομαι ιδιαίτερα, είναι και τιμή και χαρά που είμαι σήμερα εδώ στην Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων για πρώτη φορά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ως πρώτος Υπουργός από την Προεδρία της Αυστρίας. Χαίρομαι λοιπόν που μπορώ να σας ενημερώσω και για να κάνουμε και συζητήσεις για τα θέματα. Είναι η τρίτη φορά που η Αυστρία έχει την ευκαιρία να λάβει την Προεδρία της Ένωσης και είμαστε πεπισμένοι ότι και μπορούμε και πραγματικά θα καταφέρουμε από κοινού μαζί σας να προωθήσουμε πολλές νομοθετικές πρωτοβουλίες στο προσεχές εξάμεινο της Προεδρίας μας και να τις ολοκληρώσουμε. Αρχικά θέλω να ευχαριστήσω την Βουλγαρική Προεδρία οι οποίοι κατά το πρώτο εξάμεινο του τρέχοντος έτους προώθησε πολλά θέματα με θετικό τρόπο και ορισμένα ε, κατάφερε μάλιστα να τα κλείσει. Τους επόμενους έξι μήνες λοιπόν θα έχουμε τέσσερα βασικά σημεία στον τομέα των οικονομικο νομισματικών. Τον έναν τον ανέφερε ήδη ο Πρόεδρος. Θα κάνουμε κάθε προσπάθεια για την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης. Θέλουμε να επιτευχθούν σημαντικές πρόοδοι. Σε σχέση με αυτό, θα ασχοληθούμε και με την Ένωση Κέφαλη Αγορών για να την ε, προχωρήσουμε όσο μπορούμε. Δεύτερο κέντρο βάρους, η περαιτέρω εμβάθυνση της ΟΝΕ με βάση την πρόταση της Κομισιόν, τρίτη προτεραιότητα, μία πιο αποτελεσματική και πιο δίκαιη φορολογία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και τέταρτον, που είναι και αυτό πολύ σημαντικό, είναι ο προϋπολογισμός φυσικά του 19 της Ένωσης. Πρέπει να ολοκληρωθεί επιτυχώς η συμφωνία από αυτού. Τώρα να κάνω μια επισκόπηση από την πλευρά μας για την ε, σημερινή οικονομική συγκυρία στην Ευρώπη. Ως Αυστρία, κατά τη διάρκεια της ε, Προεδρίας, τώρα βλέπουμε ότι είναι καλή η ευρωπαϊκή κατάσταση, ιδιαίτερα ε, ρωμαλαία οικονομική ανάπτυξη και η κατάσταση το 2017 ήταν πολύ υψηλή όσον αφορά την ε, αύξηση του ΑΕΠ και των μεμονωμένων χωρών και της Ευρωζώνης και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε ούτως ώστε να ληφθούν μέτρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να υπάρξει μια σταθεροποίηση και τελικά μια διάρκεια αυτών των εξελίξεων. Τα τελευταία χρόνια εργαζόμενοι από κοινού επιτύχαμε να αντιμετωπίσουμε τη δυσχερή οικονομικό-πιστωτική κρίση και με αυτό τον τρόπο επανήλθε καλύτερη κατάσταση και στην αγορά εργασίας. Και αντιμετωπίστηκε και το θέμα της υπερχρέωσης των κρατών και των ελλημάτων. Είναι πολύ καλύτερη τώρα η κατάσταση. Άρα και από αυτή την άποψη είναι πολύ θετικό αυτό που διαπιστώνουμε. Σε όλα τα κράτη της Ένωσης, επειδή έγιναν και σαφείς ε, μεταρρυθμίσεις, υπήρξε αυτή η σταθεροποίηση, αυτή η θετική εξέλιξη. Τώρα μεταρρυθμίσεις. Διαπιστώνω παρόλα αυτά ότι έχουμε ακόμη ουσιώδεις προκλήσεις ενώπιόν μας. για παράδειγμα το δημόσιο και ιδιωτικό χρέος, πρέπει να αντιμετωπιστεί με περισσότερα μέτρα. Είπα ότι έχει μειωθεί η ανεργία, αλλά παρόλα αυτά σε αρκετές χώρες της Ευρώπης, ιδιαίτερη ανεργία των νέων, κατά την άποψή μας, είναι ακόμη υπερβολική. Ιδιαίτερα Οι τράπεζες αντιμετωπίζουν ε, πολλά μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Πρέπει να βελτιωθεί η κατάσταση εδώ. Παράλληλα, πρέπει να έχουμε πλήρη συνείδηση ότι η ανάπτυξη ναι μεν ε, πάει καλά αλλά δεν μπορεί να θεωρηθεί πανάκια για όλα πρέπει και η νομισματική πολιτική οπωσδήποτε να βοηθήσει μέσω μέτρων που θα μας οδηγήσουν σε μια συνεχή ανάπτυξη για την Ένωση. Ξέρουμε ότι σε διεθνές επίπεδο υπάρχουν πολλές εντάσεις. Ξέρουμε ότι ακούγονται πολλά για παγκόσμιο εμπορικό πόλεμο. Υπάρχει αυξανόμενος προστατευτισμός σε παγκόσμιο επίπεδο. Είναι σαφές αυτό. Και θεωρούμε ότι όλα αυτά είναι και ευκαιρίες και ε, προκλήσεις όμως. Και αναφέρομαι συγκεκριμένα στις ε, ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις. Και σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουμε και μια δημογραφική αλλαγή. Οπότε και εδώ πρέπει από κοινού, τώρα ακριβώς, αξιοποιώντας ε, την θετική συγκυρία, να ασχοληθούμε και με αυτά τα θέματα και εδώ να λάβουμε μέτρα, να αξιοποιήσουμε την ευκαιρία. Συγκεκριμένα, Ξέρετε ότι υπήρχε ε, στις αρχές του χρόνου συνάντηση της Παγκόσμιας Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου όπου υπόθηκε όταν λάμπει ο ήλιος είναι κατάλληλη στιγμή να φτιάξεις τη σκεπή. Αυτό νομίζω ισχύει ιδιαίτερα και για την Ευρώπη. Τώρα, για τα θέματα που θα μας απασχολήσουν ε, σε σχέση με τις αρμοδιότητές σας. Το σημαντικό θέμα είναι η Τραπεζική Ένωση. Το πιο σημαντικό. Εδώ θα εστιάσουμε. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για τη μείωση των κινδύνων και θα προχωρήσουμε κατόπιν με τη σωστή ε, ταξινόμηση και στο θέμα της ε, κατανομής των κινδύνων. Έχουμε τον οδικό χάρτη, όπου ακριβώς υιοθετείται αυτή η σταδιακή προσέγγιση, βήμα το βήμα. Και εδώ, με βάση τα πορίσματα του Συμβουλίου, Έχουμε λοιπόν αυτό τον οδικό χάρτη για να ξεκινήσουμε πολιτικές διαπραγματεύσεις για ένα, σύστημα, ένα ευρωπαϊκό σύστημα εγγύησης των καταθέσεων. Θα προχωρήσουμε σε ενέργειες γι' αυτό, αλλά πάνω απ' όλα το κέντρο της προσοχής μας θα είναι περαιτέρω μέτρα για τη μείωση των κινδύνων. Χαιρετίζω ότι έχουν ήδη ξεκινήσει τριμερείς διάλογοι για στο λεγόμενο τραπεζικό πακέτο, όπου αναφέρεται και η μείωση των κινδύνων. Και μάλιστα ε, θεωρείται ε, και από τα δύο θεσμικά όργανα πρώτη προτεραιότητα. Πρέπει λοιπόν επικοδομητικά να επιχειρήσουμε να αποφασιστεί αυτό το πακέτο πριν από το τέλος του χρόνου. Άλλη προτεραιότητα στον τομέα αυτό είναι οπωσδήποτε το θέμα των μη εξυπηρετουμένων δανείων. Πρέπει οπωσδήποτε να αντιμετωπίσουμε και να αποτρέψουμε τη δημιουργία νέων. Θα υπάρξουν νομοθετικές ε, προτάσεις κατά το εξάμεινό μας για τα θέματα αυτά. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να δώσουμε προτεραιότητα και για τον κοινό μηχανισμό ασφαλείας στα πλαίσια της δραστηριότητα του ενιαίου μηχανισμού εξυγίανσης. Αυτό το λιγόμενο Common Backstop. Τον Ιούνιο, ακριβώς στη συνάντηση κορυφής του Euro, συμφωνήσαμε ότι αυτό το Backstop θα πρέπει να προετοιμαστεί και από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό ε, Σταθερότητας. Το ESM Θεωρούμε λοιπόν ότι θα αποτελέσει και αυτό μία επιτυχία της Προεδρίας μας. Ότι μπορεί να αποτελέσει τουλάχιστον. Τέλος, για την Τραπεζική Ένωση, ένα θέμα που είναι πολύ ψηλού κόστους ε, για τις ε, διαμεθοριακές ε, συναλλαγές στο στο χώρο του ευρώ. Θέλουμε να κλείσουμε το θέμα αυτό λοιπόν κατά την Προεδρία μας. Η Ένωση των Κεφαλαίων Αγορών. Και αυτή σημαντικό θέμα. Γιατί έτσι θα εμβαθύνουμε την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα των κεφαλαίων όπου θέλουμε να έχουμε ε, αξιόπιστα ε, μέσα. Θέλουμε να υπάρχει μια πολλαπλότητα πηγών χρηματοδότησης και μία βελτίωση της πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και να επιτρέψουμε και νέα επιχειρηματικά μοντέλα. Θεωρούμε ότι θα είναι δυνατό μέσω του κανονισμού για τις ευρωπαϊκές υποδομές των αγορών, το λεγόμενο EMIR REFIT, να βοηθήσουμε τους ε, μικροεπιχειρηματίες, ιδιαίτερα στον τομέα των παραγόγων για τους κεντρικούς αντισυμβαλωμένους και θεωρούμε να προωθήσουμε και τα προϊόντα συντάξεων, τα λεγόμενα PEP. E και αυτά θέλουμε να τα, να τα προωθήσουμε. Γιατί πιστεύουμε ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε υγιή ανταγωνισμό μεταξύ των συνταξιοδοτικών ταμείων ευρέως στην Ένωση και να οδηγήσει αυτό σε εξοικονομήσεις για να έχουμε μακροχρόνιες επενδύσεις. Στη συζήτηση μαζί σας κυρίως θα ασχοληθούμε και με την ποιότητα της εφαρμογής αυτών των μέτρων. Εξίσου αναγκαία είναι να μπορεί να υπάρχει ε, διαμεθοριακή λειτουργία των επενδυτικών ταμείων και αυτό θα είναι στο επίκεντρο της προσοχής μας. Ο συντονισμός των οικονομικών πολιτικών είναι επίσης ένα θέμα που θα μας απασχολήσει κυρίως ο τομέας της σταθερότητας και της σύγκλησης των οικονομιών των κρατών μελών. Θέλουμε να τηρείται το σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης. Να το διασφαλίσουμε αυτό. Και οι συστάσεις που γίνονται στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου να τηρούνται, ούτω ώστε να έχουμε μια καλύτερη εφαρμογή και των αναχώρα συστάσεων. Η Προεδρία μας θα ε, ξεκινήσει και το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο για το 2019. Θα έχουμε τις, αιτήσει ε, τις εκθέσεις ανάπτυξης, ε, τις εκθέσεις για τους μηχανισμούς προειδοποίησης και θα κάνουμε τις απαραίτητες συστάσεις στην Ευρωζώνη για να ληφθούν αποφάσεις. Και επίσης θα στηρίξουμε τις προτάσεις των κρατών μελών για την εφαρμογή των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων. Και κυρίως θα ασχοληθούμε με την πρόταση που ήδη συζητείται στα πλαίσια του τριμερούς διαλόγου που αφορά την αύξηση των ε, πιστώσεων για την τεχνική στήριξη των μεταρρυθμίσεων. Θα εμείνουμε σε αυτό. Υπάρχει μια προσωρινή συμφωνία από ό,τι έμαθα, από τη σημερινή συζήτηση στον τριμερή διάλογο και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, ούτω ώστε έγκαιρα και κατάλληλα να καταλήξει και το θέμα αυτό. Η πρόταση της Επιτροπής για τη στήριξη των διαθροτικών μεταρρυθμίσεων θα εξεταστεί και θα στηρίξουμε τις θεσμικές και διοικητικές μεταρρυθμίσεις για να έχουμε περισσότερα αποτελέσματα. Για τη φορολόγηση. Θέλουμε περισσότερη αποτελεσματικότητα και δικαιοσύνη. Θα κάνουμε κάθε προσπάθεια για να υπάρχει διαφάνεια των φορολογικών συστημάτων να διασφαλιστεί η δημοσιονομική βάση των κρατών μελών δηλαδή να ληφθούν τα μέτρα ούτω ώστε να αποφευθεί ο επιζήμιος φορολογικός ανταγωνισμός μεταξύ των κρατών μελών αλλά κυρίως να αποφύγουμε τη φόρο απάτη και την φοροδιαφυγή. Σημαντικό θα είναι και έχει να κάνει και με την παγκοσμιοποίηση και επειδή έχει να κάνει και με τις νέες τεχνολογίες σημαντικό λοιπόν είναι να υπάρξει εξυγχρονισμός και των φορολογικών διατάξεων. Βασική προτεραιότητα για το θέμα αυτό, για την Προεδρία μας, θα είναι το θέμα της φορολόγησης της ψηφιακής οικονομίας. υπέβαλε την πρότασή της η Κομισιόν τέλη Μαρτίου επ' αυτού, ούτως ώστε οι, οι ψηφιακές πλατφόρμες να παρακολουθούνται καλύτερα. Υπάρχουν προτάσεις και του ΟΣΑ γι' αυτό και υπάρχουν και προτάσεις για την ε, φορολόγηση ακριβώς των κερδών. Την προηγούμενη εβδομάδα ε, ως πρώτο βήμα έγινε μια υψηλού επίπεδου ε, διάσκεψη στη Βιέννη, ένα πρώτο βήμα για την φορολόγηση της ψηφιακής οικονομίας. Δεν υπάρχει από αυτού τελική θέση του Συμβουλίου, θα το προωθήσουμε περαιτέρω, αλλά και το άτυπο ECOFIN στις αρχές Σεπτεμβρίου θα το αξιοποιήσουμε για να υπάρξει ε, πρόοδο αυτό. Ο εξυγχρονισμό του ΦΠΑ και κυρίω η απλούστευσή του για τι μικρομεσαίες επιχειρήσει και μέτρα για την καταπολέμηση των φοροαπατών, όλα αυτά επίση θα τα προωθήσουμε. Επιπλέον, θέλουμε και μία κοινή βάση μέτρησης του εταιρικού φόρου. Και αυτό είναι προτεραιότητα της Προεδρίας μας και θα επιχειρήσουμε να έχουμε την πιο ευρία δυνατή, το πιο ευρύ δυνατό ορισμό αυτής της κοινή ε, ε, βάσης εταιρική φορολόγησης για να υπάρχει δικαιοσύνη σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε τελευταία ανάλυση, έχει σημασία να εξετάσουμε τον κατάλογο των χωρών που δεν συνεργάζονται για φορολογικά θέματα. Αυτή είναι μια αναγκαία λειτουργική βάση για να αποφύγουμε τις φοροαπάτες και, φορο... και τη φοροδιαφυγή. Ήδη τώρα βλέπουμε ότι ο κατάλογος αυτός έχει παίξει θετικό ρόλο. Πολλές χώρες παντού στον κόσμο συμφωνούν με αυτό το πρότυπο αλλά με ιδιαίτερα πρωτοβουλιακό τρόπο θα αξιοποιήσουμε αυτό το μέσο σε παγκόσμιο τρόπο για να επιτύχουμε. Σε ό,τι αφορά τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό για το 2019, αφενός ε, έχουμε να κοιτάξουμε το ε, σχέδιο προπολογισμού του 2018 σε ό,τι αφορά και τις γενικές αρχές που ακολουθήθηκαν και σε ό,τι αφορά το θέμα αυτό θα διαθέσουμε τα απαραίτητα μέσα προς την ε, υποστήριξη των προτεραιοτήτων που έχουμε θέσει. Αυτό δε που είναι σημαντικό για την διαπραγμάτευση για το 2019 είναι να κοιτάξουμε και τις ε, κατευθυντήριες γραμμές ε, του ECOFIN του Φεβρουαρίου του 2018 και όσα αποφασίστηκαν εκεί. Προκειμένου να ακολουθήσουμε αυτή τη γραμμή στις διαπραγματεύσεις, λοιπόν. Αύριο έχουμε τον πρώτο γύρο τριμερών διαλόγων, όπου θα έχουμε και την ευκαιρία να ακούσουμε και την τοποθέτηση και να δούμε και την τοποθέτηση του Συμβουλίου σε ό,τι αφορά το σχέδιο προϋπολογισμού. Αναμένουμε και την ε, τοποθέτηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το Σεπτέμβριο προκειμένου να συζητήσουμε όλα αυτά για να βρούμε μια κοινή φορολογική, μια κοινή βάση για τον προπολογισμό. Τέλος, χαιρόμαστε που έχουμε τη χαρά και την τιμή στην τρίτη μας αυτή προεδρία να συζητήσουμε και να πραγματευτούμε πολλά θέματα σε ό,τι αφορά και τους όρους πλαίσιο που φυσικά έχουν σημασία, όπως για παράδειγμα τις διαπραγματεύσεις για το Brexit. Έχουμε και ασφαλώς ε, τις ευρωεκλογέ ε, του χρόνου και αντιλαμβανόμαστε την ευθύνη που έχουμε για να καταφέρουμε στην Προεδρία μας να ολοκληρώσουμε όσο πιο πολλά ζητήματα γίνεται και προσβλέπω στη συνεργασία μας ε, τους επόμενους μήνες σε μια κοινή επικοδομητική λοιπόν πορεία και καλή συνεργασία. Σας ευχαριστώ. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ για την πολύ Καλή αυτή η παρουσίαση και τώρα να ξεκινήσουμε με τις παρεμβάσεις των μελών. Ο Ότμαρ Κάρας είναι ο πρώτος ομιλητής. Ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ, συνάδελφοι, χαίρομαι που σας καλωσορίζω καταρχάς εδώ στην Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσίασή σας και βρισκόμαστε σε μια ιδιαίτερη κατάσταση σήμερα. Ο επικεφαλής της πρώτης ομάδας είναι όλο το απόγευμα εδώ μαζί μας και παρακολουθεί τις εργασίες μας. Ε, καλώς ορίσατε λοιπόν και υποστηρίζουμε και εμείς αυτές τις προτεραιότητες που έθεσε η Αυστριακή Προεδρία και καλώς ορίζω ιδιαίτερα την προσέγγιση για την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης. Εδώ δεν μιλάμε λοιπόν μόνο για τα θέματα ε, ΕΔΙΣ, αλλά και τα θέματα μείωση του κινδύνου σε ό,τι αφορά τι αγορέ. Ε, κατά δεύτερο θέμα, σε ό,τι αφορά την Οικονομική και Νομισματική Ένωση, παρά όλε τι προσπάθειε που γίνεται, το ευρώ εξακολουθεί να παραμένει το μοναδικό νόμισμα στον κόσμο που δεν έχει κοινή δημοσιονομική πολιτική. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να το επιλύσουμε ως πρόβλημα το συντομότερο δυνατόν. Και ρωτώ λοιπόν, η Αυστριακή Προεδρία πώς τοποθετείται έναντι του, του προβλήματος αυτού όλες οι διακυβερνητικές ε, λύσεις που μπορούν ε, και αναγκαστήκαμε να ψάξουμε να βρούμε κατά τη διάρκεια της ε, κρίσης μας και η ασπίδα διάσωσης και το ταμείο, νομισματικό ταμείο και οι σχετικοί κανόνες χρειάστηκε να μετατεθούν και να γίνουν ευρωπαϊκό δίκαιο. Αυτός ο προπολογισμός λοιπόν για το ευρώ στο συνολικό προπολογισμό θα πρέπει να ενταχθεί και θα πρέπει να τροφοδοτείται από ίδια μέσα σε ό,τι αφορά και το ψηφιακό σκέλος και αυτός ο προπολογισμό ε, θα πρέπει να χρησιμοποιείται και για μη χώρους που δεν εντάσσονται στον ευρώ για το συνολικό πακέτο έχουμε μία ειδική επιτροπή σε ό,τι αφορά τα φορολογικά ζητήματα και που ασχολείται με θέματα φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής. Και θα πρέπει λοιπόν αυτά τα θέματα να τα κοιτάξουμε στην επιτροπή αυτή. Πριν από λίγες ημέρες, η υπηρεσία καθορισμού του προπολογισμού μας ε, αποκάλυψε ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουμε τις συστάσεις αναχώρα στην Αυστρία έχουμε μόνο δύο τέτοιε συστάσει και θα ήθελα να σα ρωτήσω τα αριθμιστικά τι στοιχεία αυτά στέκουν και τι θα κάνετε σε ό,τι αφορά τις ε, συστάσεις αυτές ε, στις ε, αναχώρα αυτές να εφαρμοστούν το των δυνατόν. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτές τις πρώτες ερωτήσεις. Και θα ήθελα να συμπληρώσω σε ό,τι αφορά την Τραπεζική Ένωση ότι από τη συζήτηση στο Συμβούλιο ΕΚΟΦΗΝ και στο ίδιο το Συμβούλιο θελήσαμε να ακολουθηθεί αυτή η βαθμιαία εφαρμογή σε ό,τι αφορά τον δεύτερο και τον τρίτο πυλώνα. Και Εκεί θα επικεντρωθεί αυτός ο οδικός χάρτης που ανέφερα. Αυτό είναι απαραίτητο βήμα, γιατί γνωρίζουμε ότι και στο εσωτερικό του Συμβουλίου υπάρχουν διαφορετικές ε, απόψεις για το πόσο χρειάζεται εναρμόνιση σε ό,τι αφορά την κοινή ανάληψη κινδύνων και την περιορισμό των κινδύνων. Αλλά μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πλέον βρήκαμε μια εναλλακτική μέθοδο και εναλλακτική προσέγγιση που θα μας δώσει την ευκαιρία σε πολιτικό επίπεδο τουλάχιστον να αντιμετωπίσουμε και τον τρίτο πυλώνα εδώ. Και θα συμβάλλουμε αυτά που μας αναλογούν σε ό,τι αφορά την ε, Αυστριακή Προεδρία προκειμένου να πετύχουμε μια συμφωνία στο εσωτερικό του Συμβουλίου. Έχω εμπιστοσύνη λοιπόν ότι θα γίνουν σημαντικά βήματα, μπορούν να γίνουν σημαντικά βήματα σε ό,τι αφορά τον περιορισμό, την ελαχιστοποίηση του κινδύνου και θεωρώ ότι και σε κοινοβουλευτικό επίπεδο θα μπορέσουμε να ε, εστιαστούμε εδώ. Σε ό,τι αφορά την ε, Οικονομική και Νομισματική Ένωση, η πρόταση την οποία υπέβαλε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους, περιλαμβάνει πληθώρα θεμάτων. Και στον τομέα αυτό έχουμε κάνει μια ιεράρχηση των θεμάτων που θα πρέπει να συζητήσουμε. Καταρχάς, η ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης, την οποία συζητήσαμε πριν από λίγο, σε δεύτερο επίπεδο. Η αντίληψη σε ό,τι αφορά τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητα, σε ό,τι αφορά το backstop για το ενιαίο Ταμείο Εξυγίανση, όλα αυτά να καθοριστούν και με συγκεκριμένο πλέον τρόπο. Και εδώ θεωρώ ότι υπάρχει δυνατότητα στα πλαίσια τη Προεδρία να δημορφωθούν όλα αυτά με συγκεκριμένο τρόπο. Η εξέλιξη επίση και διεύρυνση των εργαλείων για ένα Ευρωπαϊκό Οικονομικό Ταμείο Πιστεύω ότι και αυτό αποτελεί κάτι ρεαλιστικό και πιστεύουμε ότι υπάρχει δυνατότητα να μεταξελιχθεί με τέτοιο τρόπο ο Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητα. Ασφαλώ και θα χρειαστεί να γίνουν συζητήσει και πέραν από την Αυστριακή Προεδρία σε ό,τι αφορά τα γενικότερα θέματα τη δημοσιονομική ικανότητα και έχουμε εδώ πέρα διαφορετικά στοιχεία. Καταρχάς έχουμε τη μεταρρύθμιση, την προσέγγιση μεταρρύθμισης υποστήριξης, όπου λοιπόν διαπιστώνουμε ότι είναι διαφορετικές οι τοποθετήσεις στους κόλπους του Συμβουλίου σε ό,τι αφορά το κατά πόσον χρειάζεται και σε ποιο βαθμό χρειάζεται μεταρρύθμιση. Ε, έχουμε την πρόταση της Γαλλίας και της Γερμανίας σχετικά με την ανάγκη διευκρίνησης του περιεχομένου των μεταρρυθμίσεων. Σε ό,τι αφορά τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και την εφαρμογή του εξαμήνου, αυτό το ανέφερα και εισαγωγικά. Θα προσπαθήσουμε να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να βρούμε ορισμούς και να καταφέρουμε να πετύχουμε την υλοποίηση το αναφερόμενο ποσό του 2% για την Αυστρία δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω εδώ και τώρα, αλλά θα το ελέγξω και θα σας ενημερώσω. Thank you. Ευχαριστώ πολύ. Θα έχουμε διερμηνία μέχρι τις 6.30 ακριβώς. Άρα πρέπει να διαχειριστούμε πολύ καλά το χρόνο μας. Διαφορετικά πολλοί συνάδελφοι δεν θα μπορέσουν να λάβουν το λόγο. Θα ήθελα να και στείτε στα δύο λεπτά ερώτηση, τρία λεπτά απάντηση και στη συνέχεια θα ε, ομαδοποιήσουμε τις ερωτήσεις των πολιτικών ομάδων. Περβάνς Μπερές. Ευχαριστώ πολύ. Θίξατε το θέμα ε, της δημιουργίας ενός δικτύου ασφαλείας για το ε, Ευρωπαϊκό, ε, Ευρωπαϊκό Οργανισμό Εξυγίανσης. Είχαμε μία συζήτηση με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Εξυγίανσης και έγινε λόγος για ε, μία εξέλιξη η οποία δεν είναι πολλά υποσχόμενη. Δηλαδή δεν μπορεί αυτός ο μηχανισμός να μετατρέψει μετατραπεί σε ευρωπαϊκό μηχανισμό εξυγίανσης. Δεν το επιθυμεί το Συμβούλιο. Πώς μπορούμε να προωθήσουμε αυτή τη διακυβέρνηση για αυτό το δίκτυ ασφαλείας και την περίπτωση της εξυγίανσης των τραπεζών. Γιατί πρέπει να δούμε και τη στάση των εθνικών τραπεζών σε σχέση με ένα ε, ε, ευρωπαϊκό ε, ταμείο θα θέλαμε περισσότερο να έχουμε ένα όχι ένα ευρωπαϊκό νομισματικό ταμείο, αλλά ένα ταμείο σταθερότητας γιατί νομίζω ότι η έκτην αυτή που ασχολείται με τη σταθερότητα του νομίσματος στην Ευρώπη. Τα δημοσιονομικά τα θίξατε σε σχέση με την σύσταση ενός καταλόγου που αφορά την παρουσίαση και την ιεράρχηση της Προεδρίας, θα ήθελα να σας ρωτήσω κατά πόσο υπάρχει ε, εποπτεία και reporting αναχώρα. Πότε θα συνέλθουν οι ομάδες εργασίας και ποιο είναι το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμά σας για να φτάσετε σε αίσιο πέρα σε αυτό το θέμα. Για να μπορέσουμε να ξεμπλοκάρουμε μια κατάσταση, κάτι το οποίο δεν πέτυχε η Βουλγαρική Προεδρία. Σας ευχαριστώ πολύ και για αυτές τις ερωτήσεις ε, σε ό,τι αφορά το... την προσέγγιση στην διακυβέρνηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού σταθερότητα και την μεταξέλιξη του σε ένα Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο. Θα πρέπει να γνωρίσουμε ότι στις συζητήσεις και στους κόλπους του Συμβουλίου κάποιες χώρες ε, τοποθετούνται σαφέστατα ότι βάσει των κοινοβουλευτικών ρυθμίσεων της κάθε χώρας, στην ε, παρούσα φάση υπάρχει ένα μπλοκάρισμα σε ό,τι αφορά την γρήγορη αλλαγή του μοντέλου διακυβέρνησης, αλλά θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε επ' αυτού, προκειμένου και η λύση της διακυβέρνησης για ένα κοινό backstop να ανοιχτεί ω δυνατότητα για τον Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο και να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί αυτή η δυνατότητα. Αλλά πιστεύουμε ότι η λειτουργικότητα μια τέτοια λύση ε, ενό κοινού backstop και η βάση του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου και επιμένω να το τονίζω με αυτό τον όρο, γιατί αυτή η πρόταση είναι αυτή που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αυτή που συζητείται άλλωστε. Θα κάνουμε λοιπόν ως Προεδρία ό,τι περνάει από το χέρι μας προκειμένου τα θέματα αυτά να συνεχίσουν να συζητιόνται υπό τη μορφή αυτή. Σε ό,τι αφορά τώρα τη βάση αναχώρα, τις συστάσεις αναχώρα, στο θέμα αυτό έχουμε την δυνατότητα να συζητήσουμε και τη μεταξέλιξη αυτών των στοιχείων. Καταρχάς σε διμερές επίπεδο, όπου αυτό είναι απαραίτητο και θεωρώ ότι ως Αυστριακή Προεδρία θα έχουμε τη δυνατότητα προκειμένου να σημειωθεί μια μετακίνηση της πολιτικής ατμόσφαιρα στο Συμβούλιο. Δεν μπορώ να σας υποσχεθώ εδώ και τώρα, όμως το τι ακριβώς θα πετύχουμε στα πλαίσια της Προεδρίας μας. Thank you. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Κάρολιν Νάτικεγκάλ έχει τον λόγο. Ευχαριστώ και σας ευχαριστώ κύριε Υπουργέ που βρίσκεστε ε, εδώ έχω δύο ερωτήσεις. Καταρχήν, πώς, ε, μάλλον τι θέση έχει η Προεδρία σας σε σχέση με το Ταμείο Ανάκαμψης και Εξυγίανσης και τι σκέφτεστε σε σχέση με το ΕΜΙΡ και το ΡΙΦΙΤ. Ε, εμείς θέλουμε να το διαπραγματευτούμε ως κοινοβούλιο, το θεωρείτε κι εσείς επίγον και πιστεύετε ότι μπορούμε να φτάσουμε σε μια συμφωνία υπό Αυστριακή Προεδρία. Επίσης βλέπω ότι έχετε δείξει μεγάλο ενδιαφέρον στο θέμα της ψηφιοποίησης και θα ήθελα να σας επισύρω την προσοχή στο θέμα CCP όπου θα μιλήσουμε και για το θέμα ε, της κυβερνοασφάλειας, της ασφάλειας στον ε, κυβερνοχώρο και του ε, ψηφιακού εγκλήματος. Ελπίζω να υπάρξει θετική αντίδραση από πλευρά σας σε αυτό το ζήτημα. Λοιπόν, Να ξεκινήσω με τη δεύτερη ερώτηση, αν μου επιτρέπετε, γιατί είναι απόλυτη προτεραιότητά μα στον τομέα τη φορολόγηση τη ψηφιακή οικονομία. Υπάρχει ένα πολύ ευρύ φάσμα. Έχουμε τους δύο βασικούς τομείς για να υπάρχει μια τίμια και δίκαιη φορολόγηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο της ψηφιακής οικονομίας και ή δυνατόν και σε παγκόσμια, σε παγκόσμιο επίπεδο. θα πρέπει να υπάρξει μια μεταβατική φορολόγηση της ψηφιακής οικονομίας. Αλλά αυτό είναι μόνο μια προσωρινή λύση. Πρέπει να μπορέσουμε να θίξουμε και τις ε, ψηφιακές πλατφόρμες για να υπάρξει δίκαια φορολογία. Υπάρχουν ε, προσπάθειες για αυτό που προτείνεται δικαίως για παράδειγμα, ε, που έχουν να κάνουν με τα κρυπτονομίσματα και τα κρυπτοστοιχεία ενεργητικού. Έχουμε πολλές αρνητικές εμπειρίες σε διάφορες χώρες στην, ε, στην Ευρώπη. Θέλουμε οπωσδήποτε να υπάρξει ένα κανονιστικό πλαίσιο που να βοηθήσει και τις επιχειρήσεις αυτές να αναπτυχθούν και ο τομέας της ασφάλειας σε σχέση με όλα αυτά. Άρα λοιπόν και η αντιμετώπιση της ε, κυβερνοεγκληματικότητας μας απασχολεί. Όλα αυτά ανήκουν σε αυτό το πλαίσιο και πρέπει να συζητηθούν από κοινού. Και γι' αυτό στην ε, συνεδρίαση την προηγούμενη εβδομάδα της ομάδας εργασίας διαπιστώσαμε ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε αυτά τα θέματα. Τώρα, για την εξυγένση. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, ούτω ώστε στα πλαίσια της Ένωσης ε, Κεφαλαιογοράς θα προωθηθεί και αυτό. Και συγκεκριμένα το Emir Refit ελπίζουμε να καταλήξει θετικά. Έχουμε μια καλή βάση για τις καταστάσεις κινδύνου. Θεωρούμε ότι τα μέτρα μείωσης ε, του κινδύνου και καταμερισμού του κινδύνου που ανέφερα θα ολοκληρωθούν μέχρι το Δεκέμβρη. Θεωρώ ότι θα πετύχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Μόλις Σκοτ Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Παρατήρησα ότι δεν μιλήσατε για βιώσιμη χρηματοδότηση ως προτεραιότητα, αν και η ε, Επιτροπή είχε τονίσει τη σημασία αυτού του θέματος και μίλησε για συγκεκριμένα επιτεύγματα κατά την Προεδρία σας ως Χαιρόμαστε για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί και η έκθεση στην οποία είμαι συγγήτρια δείχνει ότι υπάρχει υποστήριξη από όλες τις πολιτικές ομάδες. Θα θεωρήσετε προτεραιότητα και θεωρείτε ότι θα πρέπει να γίνουν συγκεκριμένα, συγκεκριμένες δοκιμές αντοχής στις τράπεζες έτσι ώστε να φτάσουμε σε μία ε, απότερη λύση και ως προς τις αποκαλύψεις που ε, γίνονται ως προς τους κινδύνους βιωσιμότητας θα υπάρξει κάποια εξέλιξη του θέματος κατά την Προεδρία σας. Η γενική μας απάντηση είναι ότι έχουμε μια ενεργό κοινή βάση μαζί με το Υπουργείο Βιωσιμότητας στην Αυστρία ούτω ώστε να προωθούμε τα θέματα αυτά και να λαμβάνονται υπόψη. Φυσικά θα παρακολουθήσουμε με πολύ καλή θέληση το θέμα αυτό ούτως ώστε να προωθήσουμε ακριβώς τη βιώσιμη χρηματοδότηση και τη βιώσιμη γενικά οικονομία για να γίνουν περαιτέρω βήματα στο Συμβούλιο στο ΕΚΟΦΗΝ νομίζω το Μάιο είχαμε μια παρουσίαση για το θέμα αυτό και νομίζω ότι και κατά την Προεδρία μας υπάρχει κάθε δυνατότητα να συμβάλλουμε θετικά. Ευχαριστώ. Δημήτρης Παπαδημούλης. Κύριε Λέγκελ, ε, σας καλωσορίζω ε, και σημειώνω ότι ήσασταν αρκετά συγκεκριμένος στους στόχους που θέτει η Αυστριακή Προεδρία στον τομέα της αρμοδιότητάς σας. Το σημειώνω γιατί η εκπρόσωπος της Αυστριακής Προεδρίας πριν λίγες ώρες στην Επιτροπή Περιφερειακής Πολιτικής έκανε το εντελώς αντίθετο. Δεν μας είπε τίποτα για τις πολιτικές συνοχής. Θα ήθελα λοιπόν αξιοποιώντας την ευκαιρία να σας ρωτήσω συγκεκριμένα πράγματα. Ε, θέσατε το φιλόδοξο στόχο να προχωρήσουν βήματα ουσιαστικά για την ολοκλήρωση της τραπεζικής ενοποίησης και με τον τρίτο πυλώνα. Για να γίνει όμως αυτό και να φύγει το θέμα από τις ε, ευρωπαϊκές καλένδες, πρέπει η μείωση του κινδύνου μαζί με την αμοβιοποίηση του κινδύνου να πάνε παράλληλα. Πρέπει να εγκαταληφθεί το δόγμα πρώτα πρέπει να μηδενίσουμε τον κίνδυνο και μετά να αρχίσουμε να συζητούμε την αμοιβεοποίηση του κινδύνου. Πώς βλέπει η Αυστριακή Προεδρία αυτή την προσέγγιση. Το δεύτερο, υπάρχει μια πρόταση του Προέδρου του Eurogroup, του κ. Σεντένο, που λέει ότι τώρα πρέπει να ενισχύσουμε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας να τον κάνουμε ένα Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο. Χρησιμοποιήσετε και εσείς τον ίδιο όρο. Και λέει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι αυτό πρέπει να λογοδοτεί όχι μόνο στα Εθνικά Κοινοβούλια, αλλά και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Να τον εντάξουμε στους ευρωπαϊκούς κανόνες. Όχι πια μόνο διακυβερνητική μεθόδος, αλλά και κοινοτική. Ποια είναι η θέση της Ευρωπαϊκής Προεδρίας απέναντι στην πρόταση Σεντένο. Προϋπολογισμός. Αν θέλουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία, πρέπει να μας ξεκαθαρίσετε ποιος είναι ο στόχος της Αυστριακής Προεδρίας. Θα εμείνετε στη θέση που η Αυστρία είχε ως κράτος μέλος, που λέει ότι και τα, οι πρώτες της Κομισιόν είναι πάρα πολύ γενναιόδοροι και πρέπει να περιοριστούν το ύψος του προϋπολογισμού. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βρίσκεται στην αντιδιαμετρικά αντιθέτη κατεύθυνση. Θεωρεί ότι και η πρόταση της Κομισιόν δεν είναι επαρκής. Πώς βλέπετε την ιδέα να προσθεθούν και νέοι ίδιοι οι πόροι. Και ένα τελευταίο υπάρχει τεράστια φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή, κλοπή δημοσίων εσόδων. Πώς μπορεί να προχωρήσει η εναρμόνιση κατά τη γνώμη σας για να δημιουργηθούν έσοδα και να υπάρχει και έντιμος ανταγωνισμός ανάμεσα στις επιχειρήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Βεβαίω, μου δίνει πολλή ενέργεια τι περαιτέρω συζητήσει αυτό που είπατε. Αναφερθήκατε στο θέμα του τρίτου πυλώνα τη Τραπεζική Ένωση. Βεβαίω. Ω Προεδρία του Συμβουλίου θα φροντίσουμε να προχωρήσει η συζήτηση. Αλλά νομίζω ότι με βάση το, την άποψη του Συμβουλίου πρέπει να υπάρχει η σωστή ιεράρχηση μεταξύ ε, μείωση του κινδύνου και καταμερισμού. Χρειαζόμαστε μια ευρεία βάση. Έχουμε πολύ θετική εξέλιξη επί της ουσίας για τη μείωση των κινδύνων, για τα μέτρα μείωση των κινδύνων, ιδιαίτερα για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Έχουμε μια καλή βάση για μια κοινή συζήτηση. Και στην ανταλλαγή απόψε με το Κοινοβούλιο. Και είναι πολύ θετικό ότι οι λύσεις που ήδη αναφέρθηκαν θα μπορούσαν να επιτευχθούν μέχρι τη, μέχρι τη λήξη του έτους. Παράλληλα, ανέφερα ότι με εντολή του Συμβουλίου θα ξεκινήσουμε σε αυτό το δεύτερο εξάμεινο τη συζήτηση για τον τρίτο πυλώνα με πολιτική μορφή. Και αυτό νομίζω θα προχωρήσει. Αλλά το πιο σημαντικό είναι να ολοκληρωθεί το θέμα της μίσης των κινδύνων. Επίσης, αναφερθήκατε στον ESM και την ε, διακυβέρνησή του. Οι χώρες οι οποίες με βάση την, ομοθετή, την ομοθεσία τους ε, προβλέπουν ε, τη λογοδοσία του, ES, του ESM θα πρέπει να έχουν πιο ανοιχτή στάση για την περαιτέρω εξέλιξη του ESM. Πρόθεσή μου είναι να κάνω ό,τι μπορώ, αλλά πιστεύω ότι θα χρειαστεί ε, μακρόχρονη συζήτηση για να προχωρήσει το θέμα αυτό. Ευχαριστώ, Μπάρμπαρα Κάπελ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε και αξιότιμη κυρία Υπουργέ. Χαιρόμαστε που βρίσκεστε μαζί μας σήμερα στην Επιτροπή και προφανώς στήξατε ε, σήμερα με συγκεκριμένο τρόπο τις προτεραιότητες της Αυστριακής Προεδρίας ε, και τα θέματα που μας αφορούν στην Επιτροπή μας και που μας έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν μας απασχολούν ακόμα σήμερα και θα μας απασχολούν και στο μέλλον. Τραπεζική Ένωση ε, αποτελεί θέμα προτεραιότητα και μείωση του κινδύνου. Έχουμε λοιπόν το θέμα της μείωσης ε, του κινδύνου, το τραπεζικό πακέτο είναι στη φάση του τρομερούς διαλόγου και προφανώς ε, τα θέματα αυτά είναι κόκκινη γραμμή που διαπερνάει όλα αυτά τα θέματα. Θα ήθελα λοιπόν να μας πείτε εν συντομία ποια είναι η στάση σας και η προσέγγιση μας. θέμα MPL και το θέμα πάμε ξεπληκτωμένα δάνεια και σε ό,τι αφορά την, ε, τον, τη μείωση του κινδύνου. Τα κοινά backstop επίσης. Ακούσαμε σήμερα και την κυρία Κόνικ από την ε, το Ευρωπαϊκό Νέο Συμβούλιο Εξυγένσης. Είναι σημαντικό λοιπόν όλα αυτά τα θέματα και μας είπαν ε, ότι θα πρέπει να οριστούν τα κριτήρια για το κοινό backstop, για το μηχανισμό ασφαλείας και ότι φυσικά η άμεση ανακεφαλαιοποίηση από το ESM ε χρειάζεται και ανέφερε και ένα ποσό η κυρία Κόνικ, 60 δισεκατομμύρια ως μηχανισμό ασφάλειας. Θα θέλαμε λοιπόν να ξέρουμε πώς τοποθετείται το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τα μέτρα για την ε, τα εθνικά δημοσιονομικά. Είναι πολύ ενδιαφέρον θέμα και εδώ και χρόνια έχουμε στο 11% ή 9% σε ό,τι αφορά την εφαρμογή. Θεωρώ ότι αυτό αποτελεί ένα βασικό ζήτημα και θα θέλουμε να δούμε πιο συγκεκριμένε κατευθυντήριε γραμμέ για την υλοποίηση σε εθνικό επίπεδο και πώ μπορούν να υπάρξουν συγκεκριμένε ε, προτάσει για χώρε όπου τα ποσοστά είναι πιο χαμηλά. Και ελπίζω λοιπόν ο τριμερή διάλογο να πετύχει καλή αποτέλεσμα σε ό,τι αφορά την Ένωση Κεφαλαίου Αγορών. Ναι, το μόνο, όχι ο Πρόεδρος ε, διακόπτη, δεν έχουμε άλλο χρόνο, θα πρέπει να σταματήσετε. Έχετε ήδη θέσει τρει ερωτήσει, Νομίζω ότι αρκούν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ερωτήσεις αυτές σε ό,τι αφορά την Τραπεζική Ένωση. Όπως ε, σχολιάσατε, πιστεύω ότι έχουμε μια καλή ευκαιρία, είμαστε σε καλό δρόμο σε ό,τι αφορά τους τριμερείς διαλόγους, να ακολουθήσουμε την οδό των ε, δηλώσεων. Έχουμε το πακέτο για την μείωση του κινδύνου, πετύχαμε καλά αποτελέσματα και στη συζήτηση στο ιστορικό του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου υπάρχει μια γενικότερη κοινή γραμμή η οποία έχει διαμορφωθεί με τα ατομιακά αυτά στοιχεία τα οποία αναφέρατε και σε ό,τι αφορά την ανάγκη να τεθούν σε μία προτεραιότητα στους επόμενους ε, μήνες, σε ό,τι αφορά και τους μεμονωμένους δείκτες, προκειμένου ε, επιτέλους να έχουμε και οριστικά αποτελέσματα για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Θεωρούμε ότι επίσης ε, έχουμε μια κοινή βάση αρκετά καλή για συνεννόηση. Θα πρέπει να υπάρχουν κάποιες ευκρινήσεις προφανώς για το ποια μορφή θα πάρουν οι μεμονωμένες τιμές αναφοράς και κατά πόσο υπάρχει προθυμία για εξελίξη των τελευταίων ετών που ήταν θετικέ να διαμορφωθούν με συγκεκριμένες τιμές σε ό,τι αφορά το backstop, το μηχανισμό ασφάλειας και την ερώτηση που θέσατε. Είναι πολύ νωρίς ακόμα για να ορίσουμε ένα ποσό από πλευρά του Συμβουλίου. Είμαστε ακόμα στη φάση των συζητήσεων, των διαπραγματεύσεων και θα είναι ασφαλώς και δική μας δουλειά στα πλαίσια της Προεδρίας μας να ορίσουμε σε κάποιο βαθμό και το ύψος αυτό. Σας ευχαριστώ και έχουμε μόνο 15 λεπτά στη διαθέσή μας. Να ομοδοποιήσουμε λοιπόν τις ερωτήσεις. Ο κύριος Νίτερμαγερ καταρχάς. Ευχαριστώ πολύ και σας ευχαριστώ κύριε Υπουργέ που ήρθατε εδώ. Βλέπω ότι αφοσιώνεστε σε θέματα φορολόγησης και εγώ έχω μία ερώτηση όπως ο κύριος Κάρας σε αυτό το τομέα. Τι θα γίνει με την Επιτροπή Τάξ. Μας ε, ε, κάνει μεγάλη εντύπωση η θέση της Βουλγαρικής Προεδρίας να προσέλθει και να συζητήσει το ε, θέμα, να το συζητήσει αυτό το θέμα. Ελπίζουμε να είναι ίδια η προσέγγιση της Αυστριακής Προεδρίας. Θα ήθελα επιβεβαίωση. Δεύτερον, μιλήσατε για το CCTB και τη μεταρρύθμιση του ΦΠΑ. Ε, από ό,τι Καταλαβαίνω θα το προωθήσετε, αλλά μας το αναφέρατε πολύ αφηρημένα. Δεν έχουμε ορατά αποτελέσματα. Πώς θα άρετε αυτό το αδιέξοδο και επίσης μπορείτε να προβλέψετε την ενισχυμένη συνεργασία επί του θέματος. Πολ Τάγκ. Ευχαριστώ. Σας καλωσορίζω κύριε Λέγκερ το θέμα και το δικό μου αφορά τη φορολόγηση. Έχετε μία μοναδική προεδρία, ε, ευκαιρία συγγνώμη, κατά την προεδρία σας να προωθήσετε το θέμα της φορολόγησης και ελπίζω η προεδρία σας να κάνει τη διαφορά. Λοιπόν, τώρα μία ερώτηση ως προς τον φόρο ε, ψηφιακής οικονομίας. Ε, βλέπετε μία ε, βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη λύση. Θα θέλαμε να υπάρξει ένας ορισμός της ψηφιακής παρουσίας που να συμπληρώνει τον παρόντα ορισμό σε σχέση με τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις που λειτουργούν σε αυτό το τομέα. Δεν θα πρέπει να έχουμε όχι μόνο μία χρόνια, αλλά και μακροχρόνια λύση εάν φτάσουμε σε μία βασική ε, διορ... καλώς διαρθρωμένη επίλυση του ζητήματος. Νομίζω ότι μπορείτε να απαντήσετε, κύριε Υπουργέ, για τα θέματα φορολόγησης που απασχόλησαν όλους. Σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις. Σε ό,τι αφορά την Επιτροπή Τάξε, για να απαντήσω κατευθείαν σε αυτά που με ρωτήσατε. Και στην Επιτροπή Οίκων, πιστεύω, υπάρχει δυνατότητα να συζητήσουμε τέτοια θέματα. Αλλά ασφαλώς ε, και ευχαριστώ θα συζητήσουμε και πιο επισταμένως με τον κύριο Κάρας ποια θέματα μπορούμε να συζητήσουμε πιο σε βάθος στις διάφορες επιτροπές ε, και να βρούμε μία λύση. Σε ό,τι αφορά την κοινή ευρωπαϊκή φορολογική βάση τώρα, ξέρουμε ότι το θέμα αυτό συζητιέται εδώ και πολύ καιρό αλλά πιστεύουμε ότι υπάρχει η δυνατότητα μέσω εντατικών διαπραγματεύσεων να σημειώσουμε σημαντική πρόοδο τους επόμενους μήνες και συνειδητά το θέσαμε αυτό ως προτεραιότητα της Προεδρίας μας, γιατί στον τομέα αυτό πιστεύουμε ότι η κοινή ευρωπαϊκή φορολογική βάση μπορεί να προωθηθεί και να πετύχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Αυτό το παράθυρο ευκαιρίας το οποίο αναφέρατε, την ευκαιρία που έχουμε στην παρούσα χρονική στιγμή να βρούμε κάποιες ρεαλιστικές λύσεις για το μέλλον. Πιστεύουμε ότι ακριβώς υπάρχει αυτό το θετικό κίνητρο σε πολλά ζητήματα. Η ψηφιακή παρουσία. Την ανέφερα. Το θέμα αυτό υπάρχει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και θα το επεξεργαστούμε κατά τη διάρκεια της ε, Προεδρία μας προκειμένου να πετύχουμε και καλή αποτελέσματα και σε επίπεδο ΑΣΑ και σε επίπεδο υψηλό, υψηλών αξιωματούχων στη Βιέννη παραβρέθηκαν και εκπρόσωποι του ΩΣΑ και νομίζω ότι και σε εθνικό επίπεδο μπορούμε να ξεκινήσουμε να θέτουμε και να καθορίζουμε όρους και ορισμούς που θα περάσουν και σε πιο ε, παγκόσμιο επίπεδο σε ό,τι αφορά τις υπηρεσίες τώρα. Ναι, ελπίζω να καταφέρουμε να βρούμε μια συνένεση στο δεύτερο ήμιση του έτους στα πλαίσια του Συμβουλίου, αλλά παράλληλα θα πρέπει να είμαστε και προσεκτικοί σε ό,τι αφορά αυτή τη μεταβατική φορολόγηση για να μην προκαταβάλουμε τις μελλοντικές συζητήσεις για τον ε, μελλοντικό φορολογικό συντελεστή. Κύριε Υπουργέ, στην ε, αρχή της εισήγησής σας μιλήσατε για τον προστατευτισμό και τους εμπλεκόμενους κινδύνους. Πώς θα ανταποκριθεί η Αυστριακή Προεδρία, πώς θα παραμείνει η Ευρωπαϊκή Ένωση ενωμένη και ε, ποιο είναι το σχέδιο σας για τις διαπραγματεύσεις με τους εμπορικούς εταίρους. Σε σχέση με το μέλλον της ΟΝΕ, θα ήθελα να μας πείτε για την δημοσιονομική μας ικανότητα. Όπως ε, ρώτησε και ο, ρώτησε και ο Ότμαρ Κάρας, ποια είναι η εμβέλεια της δημοσιονομικής ικανότητας, πώς μπορεί να χρηματοδοτηθεί, ποιοι θα είναι οι πόροι και από πού θα προέρχονται και τι προβλέπετε για τις χώρες που δεν βρίσκονται στην Ευρωζώνη, αλλά που έχουν δεσμευτεί να προχωρήσουν τη στιγμή που πληρούν τα κριτήρια. Άλφρεντ Σαντ. Κύριε Υπουργέ, στο πρόγραμμα της Αυστριακής Προεδρίας φαίνεται ότι είσαστε πιο φιλόδοξοι σε σχέση με την Τραπεζική Ένωση. Θεωρείτε ότι η πρόοδος είναι ένα πρόκριμα έτσι ώστε ένα πρόκριμα και προαπαιτούμενο για τον επιμερισμό των κινδύνων. Ο Μάριο Ντράγκη τόνισε ότι ο επιμερισμός ε, του κινδύνου μπορεί να ισχύσει διότι έχουμε ανταποκριθεί, στα προαπαιτούμενα. Θεωρείτε ότι αυτή η μείωση κινδύνου ίσως υποσκάπτει την αλληλεγγύη στην Ευρωζώνη γιατί πολλά εξαρτώνται από τα εμπορικά πλεονάσματα που προέρχονται από ορισμένε χώρες και γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να ξέρουμε ποια είναι η θέση της Αυστριακής Προεδρίας γιατί η κυβέρνηση Τραμπ, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, θα επιτεθεί κατά των ευρωπαϊκών οικονομιών εξαιτίας των εμπορικών τους πλεονασμάτων, γιατί η μείωση του κινδύνου είναι προαπαιτούμενο. Η τελευταία οικονομική αποτίμηση δείχνει ότι στην Ευρωζώνη υπάρχει ανάπτυξη διασυνοριακά. Αυτό έχει και αρνητικές συνέπειες. Τα στοιχεία της Eurostat δείχνουν ότι οι τιμές έχουν ανέλθει κατά 4,5% το πρώτο τρίμηνο του 2018. Ε, Δεν έχει νόημα λοιπόν να μιλάμε για λιτότητα έτσι ώστε να μην βοηθήσουμε τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους. Θεωρείται ότι τα νέα μέτρα ανάπτυξης χρειάζονται έτσι ώστε να αυξηθεί η αγοραστική δύναμη των πολιτών. Ε, έχουμε και μία σύντομη ερώτηση από τον Σβέν, στα πλαίσια του Καρστεάη. Πολύ σύντομα, μία ερώτηση για την υποχρέωση των μεγάλων επιχειρήσεων να υποβάλουν ε, δημόσιες δηλώσεις ε, για τη δραστηριότητα και, και την φορολόγησή τους. Ξέρω ότι Έχετε κάνει διμερεί συζητήσει για το θέμα αυτό, όμω το αναλυτικό πρόγραμμά σα δεν αναφέρεται. Νομίζω ότι φυσιολογικά θα ήταν να υπάρξει μια ομάδα εργασία του Συμβουλίου επ' αυτού. Το Κοινοβούλιο στηρίζει ιδιαίτερα αυτή την πρόταση. Θα μπορούσατε να μα ανακοινώσετε λοιπόν σήμερα ότι θα δημιουργήσετε αυτή την περαιτέρω ομάδα εργασία, ούτω ώστε να αποφευθεί εντύπωση ότι η θέση της ε, Αυστρικής Δημοκρατίας με, που είναι κατά αυτής της πρότασης, συγχαίρεται με το ρόλο το δικό σας που ως πρόεδρος του Συμβουλίου πρέπει να είστε ουδέτερος. Μάλιστα, να απαντήσω σε ερωτήσεις. Για το λεγόμενο προστατευτισμό, στα πλαίσια μιας, ενός κοινού μετόπου, το συνδέω και με την ερώτηση που έγινε μετά για μια κοινή στάση έναντι των ε, εμπορικών πλεονασμάτων και τις επιθέσεις των ΗΠΑ. Είπα στην εισαγωγική μου ομιλία ότι είμαστε σε φάση που είναι ιδιαίτερα απαιτητική. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε πολλές προκλήσεις, εμπορική πόλεμη, προστατευτισμός. Υπάρχει μια κάποια κλιμάκωση αυτών των φαινομένων. Το λέω ε, ευθύς εξ αρχής. Δεν έχει το ΕΚΟΦΗΝ καμία απευθύς αρμοδιότητα για τα εμπορικά αυτά θέματα αλλά με, μας ανησυχούν φυσικά, γιατί έχουν φυσικά επιπτώσεις στην συνολική ανάπτυξη και εξελίξη στην Ευρώπη. Και πιστεύω ότι η ενότητα που έχει υπάρξει στις διαπραγματεύσεις μέχρι τώρα, ότι θα διατηρηθεί, ότι θα διατηρήσουμε την κοινή μας γραμμή σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τώρα, για την δημοσιονομική ικανότητα και τι βάση θα έχει. Για μας ε, το πρώτο είναι να ευαθυνθεί η ΟΝΕ με βάση την πρόταση της Κομισιόν για τα θέματα αυτά, η περαιτέρω εξέλιξη του ESM. Βλέπουμε πολλές δυνατότητε εδώ και θέλουμε να προχωρήσουν οι συζητήσεις, να γίνουν τα πρώτα βήματα προς αυτή την κατεύθυνση και κατόπιν να συζητήσουμε και την περαιτέρω οικοδόμηση του οργανισμού αυτού. Βλέπω την πρόταση της Γαλλίας και της Γερμανίας. Θεωρώ ότι είναι καλή για να υπάρξει σταθερότητα. Αλλά πρέπει να διευκρινιστεί η συζήτηση σε επίπεδο Συμβουλίου. Πρέπει να καταλάβουμε όλοι τι επιπτώσεις θα έχει. Για την Τραπεζική Ένωση να τονίσω για άλλη μια φορά, γιατί αναφέρθηκε το θέμα της αλληλεγγύης, θεωρώ ότι πάει θετικά η συζήτηση. Βεβαίως, πρέπει να υπάρξουν μέτρα για την αλληλεγγύη, ούτως ώστε ο πυλώνας 2 να διευκρινιστεί. Βεβαίως, είπα ότι πάνε καλά τα πράγματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε διάφορους τομείς που αφορά τη βελτίωση κάποιων δικτών, αλλά σίγουρα υπάρχει ανάγκη περαιτέρω διευκρίνησης αυτών των δικτών και της ε, βάσης μέτρησης. Και τονίζω ότι δεν καταλαβαίνω την θέση μου ως ε, προεδρεύοντος, ως εκπροσώπου της Αυστρίας. Όχι. Εγώ είμαι μεσολαβητής, ούτω ώστε να προχωρήσει η ε, συνένεση και με το Κοινοβούλιο. Τώρα για τις ε, συστάσεις αναχώρα, όχι δεν είναι η δική μας χώρα, η δική μας θέση που θέλω να προωθήσουμε. Όπως προβλέπει η ε, εξέλιξη του θέματος, προσπαθούμε βήμα το βήμα να καταλήξουμε σε κοινή θέση, γνωρίζοντας ότι για τα θέματα αναχώρα είναι σημαντικό να ξεπεράσουμε και το ευρωπαϊκό επίπεδο, να συνεργαστούμε με τον ΟΣΑ και με άλλους εταίρους μας παντού στον κόσμο. Όλα αυτά θα τα προωθήσουμε ούτως ώστε να έχουμε δυνατότητα, όπως και τώρα, να ε, παρέχονται και αναχώρατα στοιχεία. Θα υπάρξει μια ομάδα εργασίας για το θέμα αυτό του Συμβουλίου. Η τελευταία ομάδα εργασίας συνεδρίασε για τον, τον Ιούνιο για το θέμα αυτό και από τα αποτελέσματα αυτά θα ε, μας βοηθήσουν να καθορίσουμε τα περαιτέρω βήματα. Ευχαριστώ πολύ για την ανταλλαγή απόψε. Ήταν πολύ χρήσιμη. Έχουμε πολύ δρόμο να διανύσουμε ακόμα και θα Ήθελα να διαβιβάσω την αίσθηση του κατεπήγοντος για να κινηθούμε σε αρκετούς τομείς. Ήταν επικοδομητική η προσέγγιση μας, αλλά θα πρέπει να προωθήσουμε τάχιστα τα όλα ζητήματα. Προτιμώ ε, να τα διαχειριζόμαστε προφορικά και όχι ε, γραπτός, όπως ε, ίσχυσε και το 2016 σε, αυτή την, ε, σε αυτό τον οδικό χάρτη. Θα θέλουμε λοιπόν να υπάρξει αυτός ο παραλληλισμός και χαίρομαι γιατί θα μας συνδράμετε και στο θέμα του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασφάλισης Καταθέσεων, το ΕΝΤΙΣ. Εάν θέλουμε λοιπόν και αυτό το backstop, θα πρέπει να είμαστε αξιόπιστοι και να μην βασιζόμαστε στην αιρεσιμότητα. Μιλάμε για ένα 8% για το backstop και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Εξυγίανσης θα βρει τα υπόλοιπα. Διαφορετικά δεν θα είμαστε αξιόπιστοι και δεν θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε από πλευράς εξυγίανσης και μηχανισμού εξυγίανσης. Γι' αυτό θα πρέπει να έχουμε και ένα αξιόπιστο μέσο στη διαθέσή μας. Τέλος, λάβαμε την ανακοίνωση για το SSM. Νομίζω ότι υπάρχουν ε, θετικά δεδομένα. Έχουμε λοιπόν τώρα μία σειρά μέτρων από πλευράς εποπτείας και βεβαίως θα πρέπει να υπάρξει και ένα συμπλήρωμα από νομοθετικής πλευράς για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Ελπίζω λοιπόν το Συμβούλιο να μας συνδράμει προς αυτή την ε, κατεύθυνση. Να δώσουμε δηλαδή προτεραιότητα στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο, λέει ο πρόεδρος. Ε, χτες ε, δεν ολοκληρώθηκε ο τριμερής διάλογος για την έδρα των δύο οργανισμών και αυτό αφορά ε, μία συγκεκριμένη εντολή για να φτάσουμε σε ένα συμβιβασμό. Έχει λήξει λοιπόν ο τριμερής και θα ήθελα να ζητήσω από το Συμβούλιο να συμφωνήσει διαφορετικά. Θα περιπλέξουμε τα πράγματα. Ξέρουμε ότι η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή έχει θέσει ε, συγκεκριμένες προθεσμίες. Είναι επίγοντο το θέμα λοιπόν και κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Τώρα εξαρτάται από το Συμβούλιο να ολοκληρώσει.